Ε. Συνάδελφοι, αν και δεν βλέπω αθρώα προσέλευση, πρέπει να ξεκινήσουμε. Περιμέναμε. Το ακαδημαϊκό τέταρτο πέρασε. Εύχομαι και ελπίζω να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. να καλωσορίσω τον Τζον Μπέλ, που είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Βιοοικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα μας ε, παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση του Food 2030. Είναι ένα project εξαιρετικά σημαντικό για την Επιτροπή μας, την DG Agri και την DG Έρευνα, που ήδη συνεργάζονται σε πολλούς τομείς για να προωθήσουν την εφαρμογισμένη έρευνα, την καινοτομία, τη γνώση την ψηφιακή οικονομία στις περιοχές της υπαίθρου. Αυτή η στρατηγική προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία στον ε, γεωργικό τομέα είναι θεμελιώδης για να εγγυηθούμε την ε, διαφοροποίηση και να συμβάλλουμε στη δημιουργία πιο βιώσιμων ε, διατροφικών συστημάτων, πιο ανθεκτικών, πιο ανταγωνιστικών, πιο υπεύθυνων και αποδοτικών. Και εύχομαι πραγματικά μετά από την εισήγηση του Διευθυντή Μπέλ να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και τώρα θα δώσω αμέσως το λόγο στον Τζον για να μας κάνει αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πάολο Ντικάστρε που έχετε παίξει πρωτοπόρο ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή Food 2030 που ξεκίνησε στο Μιλάνο στην Expo που ο Δόκτωρ Δεκάστρο και άλλοι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου συνέβαλαν στην ε, εκπόνηση μιας στρατηγικής για την ε, το σύστημα των τροφίμων και πώς το βλέπουμε από την άποψη της έρευνας και της ανάπτυξης είναι διαφέρει δική μας προοπτική από αυτό που είδατε το πρωί και τις ρυθμιστικές ε, ε, διαδικασίες. Εγώ είμαι διευθυντής της έρευνας και της καινοτομίας, εξετάζουμε τα ε, ε, σύστημα γεωργίας και τροφίμων ε, πιο μακροπρόθεσμα. Εξετάζουμε τις τάσεις, τα σημάδια ε, που προκύπτουν από την κοινωνία και προσπαθούμε να προτείνουμε λύσεις. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για το Food 2010 που είναι η πρώτη φορά που κάναμε έρευνα και καινοτομία και σχετική στρατηγική για να εξετάσουμε τις ανάγκες και τις ευκαιρίες για το σύστημα το αγροδιατροφικό μέχρι το 2030 που θα πρέπει να έχουμε καταλήξει σε μια βιώσιμη προσέγγιση. Θα μιλήσω για την έρευνα και την καινοτομία και τη σχετική πολιτική που εξετάζει τα τρόφιμα και την ασφάλεια στην ε, διατροφή όταν πρέπει δηλαδή να μετακινηθούμε σε ένα βιώσιμο σύστημα. Και τρία βασικά μηνύματα θα προσπαθήσω να σας διαβιβάσω. Το ένα είναι ότι το σύστημα το αγροδιατροφικό είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία και ω οικονομία τα επόμενα 20 περίπου χρόνια. Και δεύτερον, να σας ε, ε, εξηγήσω ότι αν και έχουμε συγκεκριμένους τομείς ε, νομοθετικούς θα πρέπει να το θεωρήσουμε όλο ένα σύστημα είτε πρόκειται για τρόφιμα από τη ξηρά είτε από τη θάλασσα που θα πρέπει να καταλήγουν στον καταναλωτή. Μια λυσίδα δηλαδή, να δούμε το δυναμικό των όσων εργάζονται στην βιομηχανία τροφίμων και αυτούς που έχουν τις πιο καινοτόμες ιδέες και πώς μπορούν όλες αυτές να ταχθούν μέσα στο ίδιο σύστημα. Τρίτη πτυχή είναι ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι με την ευρωπαϊκή πολιτική και τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν δεσμευτεί να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να θεσπίσουμε ψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας για την έρευνα και την κοινοτομία ώστε να καταλήξουμε σε λύσεις και συμπεράσματα σε αυτούς που θα πρέπει να ε, ε, τα εφαρμόσουν στην πράξη εκεί όπου ζουν και ψηφίζουν. Το θέμα της ε, συνοχής της πολιτικής προκύπτει λοιπόν για μας που κάνουμε έρευνα και κοινοτομία στην Κομισιόν. Δεν είμαστε συχνά με, μετέχοντες στην διαδικασία συναπόφασης, εμείς χρησιμοποιούμε τα προγράμματα πλαίσιο όπως το Horizon 2020, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τους συναδέλφους που οδηγούν στην απλοποίηση και εξυγχρονισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής, το πρόγραμμα πλαίσιο 9 για το μέλλον και τα επενδυτικά κονδύλια για διάφορους τομείς. Εδώ είναι ένα, σε μια διαφάνεια που δείχνει την αποκάλυψη, την τέλεια καταιγίδα. Δεν συνειδητοποιούμε συχνά ότι το σύστημα από την παραγωγή στην κατανάλωση στην ουσία βρίσκεται στην καρδιά όλων των μεταβατικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Γνωρίζουμε ότι όπως είπε και ο πρόεδρος Μακρόν, δεν υπάρχει άλλος πλανήτης. Δεν έχουμε χώρο ελιγμού ε, περιθώριο λιγμού όσον αφορά τις επιλογές και τους διαθέσιμους πόρους και τους χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Όταν υιοθετήθηκε το PDP εδώ, όταν υιοθετείται μάλλον το PDP και η Επιτροπή Προπολογισμού θα λάβει σημαντικές αποφάσεις στους επόμενους μήνες, έχουμε μόνο 10 εσοδίες για να καταφέρουμε τους στόχους που έχουμε θεσπίσει για το 2030, δηλαδή δύο θητείες του Κοινοβουλίου ή δυόμιση ε, κύκλους του προϋπολογισμού. Λίγο χρόνο έχουμε λοιπόν για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Και τι σημαίνει αυτή για τις κλιματικές αλλαγές, όπως έχετε δει από τις πρόσφατες συζητήσεις στην Βόνη, η τα διατροφικά απόβλητα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ε, ε, ρηπογόνος παράγοντας παγκοσμίως μετά από την Κίνα και τη ΣΥΠΑ. τα απόβλητα τα διατροφικά εκτός της Ένωσης και στο επίπεδο της Ένωσης όμως αποτελούν, είναι το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται. Το 1 τρίτο των τροφίμων χάνονται. Αυτό σημαίνει δηλαδή πολλά όσον αφορά τη δομή της οικονομίας της κοινωνίας μας και μόνο και μόνο με τα απόβλητα τα διατροφικά μπορούμε να κάνουμε μεγάλη αλλαγή. Επόμενη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα στο Κατοβίτσες της Πολωνίας θα εξετάζει το, το πώς μπορούμε να εργαστούμε στον τομέα της γεωργίας και στα συστήματα τροφίμων ώστε να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου. Πρόσφατα στην Ευρώπη για πρώτη φορά ε, υπήρξαν ε, κυκλώνες που και επηρέασαν την Ευρώπη και γεννήθηκαν στον Ανατολικό Ατλαντικό. Είναι η αρχή ενός νέου ε, κλιματικού φαινομένου. Είχαμε δηλαδή ε, καιρικά φαινόμενα τελείως διαφορετικά. Η Γαλλία έχασε το 1 τρίτο της ε, σοδιάς σιτηρών ε, το περασμένο χρόνο και στην Πολωνία είδαμε ότι η περίοδος ε, καλλιεργίας είναι διαφορετική ε, από χρόνο σε χρόνο και γι' αυτό έχουν δυσκολίες με τη χρήση του ύδατος ε, και εξετάζουν τα εδάφη για να δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά και πώ να εμπλουτίσουν τα εδάφη τους να δούμε τους στόχους που έχουμε όσον αφορά το διπλό στόχο της παχυσαρκίας και της ε, πείνας. Ε, εμείς έχουμε καταφέρει στο δυτικό κόσμο έχουμε, είναι, να έχουμε περισσότερους παχύσαρκους από ό,τι έχουμε πεινασμένους. Ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο έχουμε τρία δις που εξαρτώνται από την ε, αλληλεία για την διατροφή τους σε πολύ ευαίσθητα μέρη του κόσμου, όπου δηλαδή τα, τα, τα αποθέματα κινούνται, μετακινούνται περαστικά. Αλλάζουν λοιπόν ε, τα μοντέλα διατροφής ε, από την φυτοφαγία στη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες στην διατροφή. Έχουμε λοιπόν αντίκτυπο στους γείτονές μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το θέμα είναι λοιπόν πού θα βρούμε πρωτεΐνες για τα συστήματα διατροφής και τα συστήματα ζωοτροφών επίσης. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται το νερό και η ενέργεια σε συστήματα τα αγροδιατροφικά. τεράστιε αλλαγές πρέπει να γίνουν αν όντω θέλουμε να θρέψουμε τα 9 δις που θα ζουν. Με 6% αύξηση της ζήτησης, ε, μεγάλη αύξηση επίσης στην ζήτηση πρωτεΐνης, μεγάλες κλιματικές αλλαγές και ακραία πίεση, ακραία πίεση στα εδάφη, στα φυτά, στα ζωντανά, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων. Αν ταυτόχρονα δούμε τα οικοσυστήματα όπου όλα αυτά γίνονται, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στην βιοπικιλότητα σε διάφορα είδη και σε διαφορετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε ακόμα συστηματικά, αλλά πάντως υπάρχουν βασικά αλλαγέ στα σχήματα της βιοπικιλότητας στην γη αλλά και στους ωκεανούς. Κάτι ακόμα, καθώς θα κάνω αυτή την παρουσίαση και θα μιλάμε για τα διατροφικά συστήματα, μιλάμε για τη γη και για τη θάλασσα. Και εκεί υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δύο. Δεν θα λύσουμε λοιπόν πολλά από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάνοντας αλλαγές διαφορετικές σε διάφορους τομείς. Χρειάζεται μια συστημική συνολική προσέγγιση που θα αλλάξει ολόκληρο το σύστημα διατροφής, τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά τα συστήματα για να τα καταφέρουμε και στο Μιλάνο, όταν, στη διάρκεια της ΕΞΠΟ, είδαμε με τον δόκτωρα Δεκάστρο ότι δεν θα υπάρξει ασφάλεια χωρίς να υπάρχει ασφάλεια των τροφίμων και δεν υπάρχει ασφάλεια των τροφίμων χωρίς ασφάλεια διατροφής και τροφίμων. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τις θερμίδες αλλά τη διατροφή. Και η ίδια συζήτηση και ξέρω έχετε ταυτόχρονα και μια μεγάλη συνεδρίαση για την Αφρική ε, αυτές τις ημέρες και θα πρέπει να φτιαχτούν συστήματα για να μπορέσουν να τα στηρίξουν όλα αυτά. Εδώ, σε αυτό το Δημοκρατικό Σώμα, είναι επίση σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα σύνολο πολιτικών ευκαιριών και πλαισίων που θα χαρακτηρίσουν τα όσα θα κάνουμε στο μέλλον. Έχουμε διάφορες λοιπόν προτεραιότητες. Είτε μιλάμε για απασχόληση, είτε για τους στόχους βιώσιμη ανάπτυξη, είτε για τους στόχους κλιματικής αλλαγής, είτε για τους στόχους του επενδυτικού, Θα πρέπει να δούμε ότι στο επίκεντρο είναι το σύστημα τροφίμων. Όποιον στόχο και αν χρησιμοποιήσουμε για το σύστημα τροφίμων απασχολεί ε, τον έναν στου πέντε πολίτε. και είδαμε το σχέδιο ανακοίνωση για την κοινή γεωργική πολιτική και αν δούμε τα νούμερα, όποιο τρόπο και από όποια πλευρά και το κοιτάξουμε, περίπου ένα στου πέντε πολίτες ασχολούνται με την γεωργία ή τη βιομηχανία τροφίμων. Ε, είναι μεγαλύτερη η βιομηχανία μας από ε, μια μισή φορά από αυτήν τον ΙΠΑ, αλλά οι επενδύσει είναι οι μισέ ε, από ό,τι στις είπα είναι η μεγαλύτερη μεταπητική βιομηχανία μας στην Ευρώπη. Τελευταία φορά όμως που ακούσατε να γίνεται λόγος για 4,5 εκατομμύρια κόσμο που εργάζεται στην ε, βιομηχανία τροφίμων στην Ευρώπη. Μόνο αν υπάρξει πρόβλημα το ακούμε πόσο μεγάλη πρόκληση είναι αυτή και καταλαβαίνετε πόσο τεράστια πρόκληση είναι αυτή για την Ευρώπη όταν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα επικρατήσουν σε μια βιομηχανία που απασχολεί τόσο πολύ κόσμο. Είναι περίσης, επίσης το 6% του ΑΕΠ μας, αλλά είναι το μεγαλύτερο μεταπητικό μας ε, ε, stand, ε, κέντρο. Αυτό που έκανε λοιπόν η Airbnb για τα ξενοδοχεία, διαφορετικά μοντέλα που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και καταναλώνεται το φαγητό. Θα πω και δύο λόγια αργότερα για το τι ακριβώς ε, βλέπουμε με τη χρηματοδότηση του προγραμματός, ε, αλλά βλέπουμε πολύ σπουδαίες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ε, καλλιεργείται, παράγεται, αξιοποιείται και δίνεται στους καταναλωτές το φαγητό. Και αυτό θα αλλάξει δραματικά τα επόμενα δέκα χρόνια. Τα τρόφιμα όλο ένα και περισσότερο θα γίνονται πιο ατομικά. Θα βασίζονται στον ατομικό βιότυπο κάθε ανθρώπου, ε, θα ε, γίνονται με ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, θα κατασκευάζονται ε, και τα συστήματα παράδοσης που θα φτιαχτούν από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα αντικατασταθούν από διαφορετικά μοντέλα, το ίδιο δυναμικά με το ότι έχει γίνει σε άλλους τομείς και πρέπει γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη. Επίσης μπορούμε να δούμε πως υπάρχουν ζητήματα σε διάφορα τμήματα του συστήματος των τροφίμων. Ας πούμε, αν κανείς οργανώνει την επιχείρησή του για τη γεωργία, θα πρέπει να έχει στοιχεία, να έχει δεδομένα. Ποιος έχει στην κατοχή του τα δεδομένα στο τομέα των τροφίμων, αυτό θα επηρεάσει τη ζωή των γεωργών στο μέλλον. Να δούμε τα μέτρα που λαμβάνονται και το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να καταφέρουμε μια βιώσιμη μετάβαση. Το πρόγραμμα Food 2030 λοιπόν είναι η προσπάθειά μας να δομήσουμε πώς θα περιχαρακώσουμε το σύστημά μας και με ποια εργαλεία έρευνας και καινοτομίας <coughs> στους όσους ασχολούνται με αυτό το τομέα. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν ένα ε, πρόγραμμα και έρευνας και τανατομίας και να εξετάσουμε λοιπόν ολόκληρο το σύστημα από την ε, παραγωγή στην κατανάλωση ε, και να δούμε τέσσερις προτεραιότητες, τέσσερις κυρίους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα συστήματα μέσω της πρόκλησης για την κλιματική αλλαγή, το θέμα της διατροφής, κυκλικότητα που σας μίλησα για τα απόβλητα νωρίτερα, που θα πρέπει να μετατραπούν σε ένα σύστημα αξίας και πώς θα μπορέσουμε με την καινοτομία να χειραφτήσουμε και κοινότητες. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε τα μέσα για μια δομημένη απάντηση ε, να την ε, ψηφιοποιηθεί με τρόπο όπως ήρθε και ο ηλεκτρισμός σε αυτούς που τον χρειάζονταν περισσότερο πριν από κάποιες ε, δεκαετίες και να μπορέσουμε να συνδέσουμε μεταξύ τους διάφορους παραμέτρους του συστήματος. Αλλά έχει να κάνει και με το χώρο, τον πραγματικό κόσμο που εργάζεται και αναπτύσσει το σύστημα. Προσπαθούμε να δούμε τον τρόπο αλληλοσύνδεσης των περιφερειών. Ας πούμε, Urban Food Policy υπήρχε στο Μιλάνο που δίνει και καλύπτει ένα σωρό αλλαγές. Έχουμε και και μια άλλη εκδήλωση στην Πολωνία αυτή την εβδομάδα για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα τοπικά συστήματα της ε, αγροτροφιμοβιομηχανίας ε, και έχουμε το PDP, το πρόγραμμα πλαίσιο, πώς αυτό θα πρέπει να ε, στηθεί, πώς θα εξυγχρονιστεί η κοινή γεωργική πολιτική, πώς θα γίνει ταυτόχρονα μεταφορά ε, γνώσης και τεχνολογίας, πώς τα επενδυτικά προγράμματα θα στοχεύουν στην πραγματική οικονομία. Οπότε, αν σύντομα δούμε μια-δυο διαφάνειες, εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα για το τι μπορεί να προσορθεί στο σύστημα. Αν δούμε κάποια από αυτά τα παραδείγματα, αυτά είναι πράγματα που ήδη έχουν ξεκινήσει ή που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος. Βλέπουμε, ας πούμε, πώς η φωτοσύνθεση, την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της φωτοσύνθεσης 1% έχουμε αποδοτικότητα, αν πάμε στο 2% θα καλύψουμε όλες τις διατροφικές ανάγκες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να γίνει. Πρέπει δηλαδή οι καλύτεροι να ασχοληθούν για να βελτιωθεί το σύστημα. Εναλλακτικέ στο κρέα, όπω λένε πολύ μεγάλο κομμάτι του συστήματο, άσχετα από το τι πιστεύουμε για τη δική μας θέση, για τα, το κρέας ή τα ζώα κτλ. Υπάρχουν τρόποι, πόροι μάλλον, που θα πρέπει να αναπτυχθούν για την ε, παραγωγή πρωτεϊνών σε άλλα διαφορετικά τρόφιμα από ότι το κρέας. Τώρα, διαφορετικοί τρόποι για τις υδατοκαλλιέργειες. Ε, ε, έχουμε διάφορα ε, μαγαζιά ή αγροκτήματα που λειτουργούν με υδατοκαλλιέργεια και ό,τι παράγεται εκεί χρησιμοποιείται για να τροφοδοτηθούν φρέσκα τρόφιμα και λαχανικά στη γειτονιά και το νερό που χρησιμοποιείται ανακυκλώνεται. Ε, ε, νέο είδος δηλαδή κυκλικών συστημάτων τροφίμων που έρχονται στις γειτονιές και υπάρχει ένα, ένα τέτοιο σύστημα ήδη στις Βρυξέλλες. Τώρα, ε, προσωποποιημένη διατροφή που μπορεί να σας φανεί πολύ παράξενο, αλλά ε, φτάνουμε σε ένα σημείο που μία από τις μεγάλες ε, επαναστάσεις ε, στην επιστήμη είναι ο βιότυπος. Καταλαβαίνουμε τα καλά βακτήρια τα οποία ε, ε, βλέπουμε ότι το κάθε, ο κάθε άνθρωπος είναι σαν ε, ένα οικοσύστημα και αν αυτό μπορούμε να το επεξεργαστούμε αρκετά μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε συμπληρώματα διατροφής ή τύπους διατροφής που θα ελέγχονται και θα συνδέονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Ας πούμε αν κανείς έχει αλλεργία στα σκυρούς καρπούς μπορεί να φτιάξει το φαγητό του σπίτι του, να τυπώσει τι χρειάζεται και χρειάζεται συγκεκριμένα συμπληρώματα και, και, αυτά μπορεί κανείς να τα τυπώσει σπίτι του. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από δυσφαγία, δεν μπορούν να καταπιούν. 50.000 ε, άνθρωποι στην Ευρώπη. Ε, ε, ε, εκεί θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για να κατασκευαστεί ένα είδος τροφής που να μπορούν να το απορροφήσουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να καταπίσουν ή πιο, ή πιο ηλικιωμένοι ή ένα σωρό ε, παθήσεις ή ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν και ένα σωρό ζητήματα που αφορούν τη διατροφή, την κατανόηση της ε, ε, διατροφής, ε, ιδιαίτερα στα ευάλωτα, σε ευάλωτες περιόδους της ζωής, πριν και μετά τη γέννηση, όταν ο κόσμος αρρωσταίνει, όταν μεγαλώνει. Και επίσης θα, πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο σε ολόκληρο την υφήλιο, πώς θα μπορούσαμε να ε, επωφεληθούμε από την αφρικανική δίαιτα, για να βρούμε δηλαδή εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να στηρίξουν ε, τα χρήματα των φορολογουμένων μας μέσω των προγραμμάτων που γίνονται ήδη. Προσπαθούμε, εδώ έχετε ένα κατάλογο από προγράμματα, προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικέ πηγές ε, τροφίμων και ζωοτροφών. Δείτε τι κάνουμε στους ωκεανούς, ελέγχουμε σε κλίμακα μακροφυκιών, δηλαδή ε, μπορούν να απορροφήσουν τα νητρικά άλατα και μπορούν μετά να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βιοπλαστικών, χημικών, καλλιτικών Έχουμε ήδη μέσω μιας πρωτοβουλίας που των 3,5 εκατομμυρίων να δούμε πώς από το σύστημα ε, των αποβλήτων μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να έχουν περισσότερα εισοδήματα οι ίδιοι ε, οι γεωργοί. Ας πούμε μπορεί ε, απλά και μόνο τα ξερά χόρτα να αποτελέσουν καύσιμο ή τα παράγωγα από την παγωγή γάλακτος μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή γίνεται μια ε, επανάσταση στη βιοοικονομία και αυτό θα καθοδηγήσει την ε, οικονομία της υπαίθρου στο μέλλον. Το θέμα είναι οι γεωργοί και οι κοινότητες θα συμμετέχουν σε αυτή την οικονομία και θα την ιδιοποιηθούν. Ελπίζω πως εμείς θα τους βοηθήσουμε να το κάνουν αυτό. Τεράστιες αλλαγές γίνονται, ακόμα και αστική γεωργία αναπτύσσεται, ιδιαίτερα στην Κίνα ε, αστική δασοπονία. Ο κόσμος ξανασκέφτεται πώς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες οι πόλεις ώστε να φέρουν την παραγωγή πρωτεϊνών μέσα στις πόλεις και βέβαια και η ψηφιοποίηση για τη σχέση με τον καταναλωτή. Πολλά γίνονται, πολλά αλλάζουν λοιπόν. Πολλές λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο το σύστημα της γεωργίας και των τροφίμων, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και επανάσταση και έχουμε στις κοινότητές μας, στην έρευνα και ανάπτυξη, στις μικρές εταιρείε και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις έχουμε μέσα για να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα αυτό δεν θα είναι ο κοιμόμενος γίγαντας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ θα πρέπει με κάθε ε, ε, ε μας ε, δύναμη να ξυπνήσουμε αυτόν τον γίγαντα. Η εργασία λοιπόν του Κοινοβουλίου από την αρχή της ΕΞΠΟ και στα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμη η εργασία εδώ, γιατί θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις ώστε να κινητοποιηθεί η έρευνα, η βιομηχανική και η γεωργική έρευνα και η έρευνα στην κοινότητα των κατασκευαστών τροφίμων για να προχωρήσουμε στο επόμενο πρόγραμμα και το επόμενο χρόνο με τη Βουλγαρική Προεδρία θα έχουμε ε, μια ε, εκδήλωση ψηλού επίπεδου στο Πλόφτη 14 και 15 Ιουνίου του 2018 <coughs> και η Αντιπρόεδρος Μαγκίνες είναι εδώ Ήσασταν εδώ από την έναρξη αυτή τη πρωτοβουλία από πέρσι. Είχαμε ισχυρή στήριξη από το Ευρωκοινοβούλιο. Η, η, η, αν δεν ξέρω αν την Παγκόσμια ημέρα τροφίμων ε, το 2018 θα θέλατε να επανέλθετε σε αυτά τα θέματα, εγώ ευχαρίστω θα έρθω να στηρίξω οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία ή να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτησή σα και να συνεργαστώ μαζί σα ώστε να εντοπίσουμε κάποιε λύσει. Όπω όλοι γνωρίζουμε, τα τρόφιμα είναι η άτυπη κοινή γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενώνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο τραπέζι λαμβάνονται περισσότερες ε, αποφάσεις που έχουν σημασία για τον κόσμο και ε, στη γεωργική κοινωνία και που εργάζονται, που ζουν, όπου θρέφονται και πώς θα μπορέσουμε να τονώσουμε την οικονομία σε ολόκληρη την Ευρώπη σε αυτό το τομέα γιατί ολόκληρη η Ευρώπη έχει μεγάλη ευκαιρία εδώ και φαντάζομαι ότι πολλά περισσότερα περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι παρά να επενδύουμε απλά χρήματα στην έρευνα και στην τεχνολογία ε, ε, και να μην τα επενδύσουμε εκεί που πραγματικά χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. Μίλησα λίγο περισσότερο από ό,τι μου είχατε πει αρχικά, αλλά ε, είμαι στη θέση σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πραγματικά ε, κύριε Διευθυντά Μπέλ για την παρουσίασή σας, για τις σημαντικές λαβές που μας δώσετε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με αυτό. Και πιστεύω πως ε, η εισήγησή σας θα μας επιτρέψει να αρχίσουμε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που το ζητούν και να πω ότι η καινοτομία δεν είναι σε αντίφαση με την παράδοση. Αν το σκεφτείτε καλά, συνάδελφοι, μπορούμε μάλιστα να πούμε πως η παράδοση σε αυτό το τομέα είναι, σε αυτόν τον αγροδιατροφικό τομέα, είναι μια καινοτομία για την έξοδο. Λοιπόν, να αρχίσουμε την συζήτηση. Ξεκινάμε με την Αντιπρόεδρο Μαρία Μαγκίνες και μετά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θέλουν. Um, Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Τζον, για την παρουσίασή σου. Με ενέπνευσε αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι η καινοτομία έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση. Συμφωνώ πλήρω. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις δραστηριότητες του προγράμματος αυτού και πιστεύω ότι αυτό που μας απασχολεί όλους εδώ είναι πώς αυτά τα πράγματα θα μεταφραστούν στην πράξη για τους παραγωγούς. Και θα ήθελα να μας δώσετε κάποια παραδείγματα ε, πραγμάτων που θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή Γεωργίας, η Επιτροπή Άγκρη, ε, έτσι ώστε αυτές οι ιδέες να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Επίσης, αυτόν τον καιρό συζητείται το θέμα της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Έχετε εξετάσει εσείς ποιες μεταρρυθμίσεις, ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να είναι σκόπιμες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Τρίτο και τελευταίο. Είναι το ερώτημα του ρόλου των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που κάνουν πολλά, υπάρχουν άλλα όμως που αδρανούν. Και το ερώτημα είναι οι γεωργοί που ενδιαφέρονται να βρουν βέλτιστες πρακτικές, πού μπορούν να τις αναζητήσουν γιατί σε κάποιους από αυτούς τους τομείς πρέπει κανείς να το δει με τα μάτια του για να πιστέψει ότι μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, στην πραγματικότητα η κύκλικη οικονομία. Και το ερώτημα που τίθεται ε, επίσης είναι εάν θα υπάρχει και οικονομική βιωσιμότητα. Εάν ακολουθήσουμε τα συμπεράσματα της έρευνάς σας καταλήγουμε σε ένα μοντέλο το οποίο να είναι και οικονομικά βιώσιμο. Ο κύριος παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, νόμιζα ότι ξεκινούμε στι 3 και όχι στι 2.30. Επομένω, ίσω να έχετε ήδη πει αυτό που σκόπευα να σα ρωτήσω. 30 εκατομμύρια τόνου σόγια ε, εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρόνο. Και ζητού, συζητούμε το ζήτημα της διατροφικής αλλαγή. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα τεράστιο κενό. Γιατί να χρειάζεται να εισάγουμε τόσο πολύ σόγια. Είναι το ζήτημα της των γενετικά μεταλλαγμένων. Ίσως χρησιμοποιώντας τα γενετικά μεταλλαγμένα οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να λοιπόν μια τεχνολογία η οποία υπάρχει και η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των τροφίμων. Θα μπορούσα να δώσω και άλλα παραδείγματα. Όμως το λόμπι των οικολόγων έχει κατατρομοκρατήσει τους πάντες και δεν ε, τη χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Εσείς προτείνετε κάποιες νέες τεχνολογίες, κάποιες ιδέες, κάποιες νέες τεχνολογίες. Αυτό που με ανησυχεί είναι μήπω πάλι η το λόμπι των οικολόγων ε, κατα, καταφέρει και δεν τις αξιοποιήσουμε γιατί οποτεδήποτε έρχεται μια ιδέα από το, τις μεγάλες εταιρείες του τομέα θεωρείται αυτομάτως κακή. Ε, thank you very much. That was a, fascinating... Ε, Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φλανάγκαν. Ε, ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσίαση, ήταν πολλές οι ιδέες. Αναφέρατε πάνω από τα τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ε, βιομηχανία των τροφίμων. Ξέρετε ακριβώς ε, τι αναλογία υπάρχει με αυτούς που ασχολούνται με τη γεωργία, γιατί αν ελέγξετε στο ίντερνετ θα δείτε διάφορα συστήματα ε, γεωργίας ε, με drones που μιλάνε ακόμα και ε, ποια θα είναι λοιπόν η θέση των ανθρώπων στη γεωργία στο μέλλον. Μίλησε, πραγματικά τι θα γίνει στο μέλλον αν θα, η κόρη μου θα με ρωτάει τι είναι ο Γιώργος τι θα της απαντώ κυρία Σέμπρα Καταρχάς, ήθελα να ρωτήσω τι έχει γίνει με τους ε, γεωργούς. Ε, πού βρίσκονται μέσα σε αυτά τα προϊόντα, σε αυτή την έρευνα. Κάθε χρόνο αναγνωρίζουμε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, αλλά έχω την αίσθηση ότι αντί να βάζουμε τους πόρους, τους ερευνητικούς σε κάτι που υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει όπως η αγροτική οικολογία, τελικά προσπαθούμε να φτιάξουμε συστήματα τα οποία μας οδηγούν όλο και περισσότερο σε μια γεωργική παραγωγή που θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την υψηλή τεχνολογία, που είναι πιο ακριβή για τους ε, γεωργούς. Θα ήμουν ευγνώμων αν μου λέγατε τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας να τους ε, εξαλείψουμε τους ε, γεωργούς. Να έχουμε μια βιομηχανία τροφίμων ή μια βιομηχανία υποκατάστατων τροφίμων. Πραγματικά, θα ήθελα να μου εξηγήσετε και ποιες είναι οι προοπτικές για την Αφρική. Είμαι μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι οι αφρικανικές χώρες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα μόνες τους να φτιάχνουν και να καλλιεργούν το φαγητό τους το να δαπανάς ε, τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων για να βρεις μια λύση για την Αφρική ενώ δεν εμπλέξεις την ίδια την Αφρική δεν έχει νομίζω νόημα. Ναι, ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο σε αυτή τη φάση, δίνω το λόγο στον Τζον Μπέλ για να απαντήσει. Α, η κυρία Πετία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση κύριε Μπέλ. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ εν συντομία να μας εξηγήσετε. Επειδή αναφερθήκατε σε όλη αυτή την έρευνα η οποία θα μας οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που κάνατε, πόσες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν κατά αυτόν τον τρόπο και σε ποιους συγκεκριμένους τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πετίβα. Ο κύριος Βαρντές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις γιατί αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή. Έχω ασχοληθεί με το θέμα, έχω ρωτήσει καθηγητές που ασχολούνται με το θέμα και δεν μιλάνε για την κλιματική αλλαγή, αλλά θέρμανση του πλανήτη, υπερθέρμανση του πλανήτη, που όταν έρθει θα έχουμε προβλήματα με πληρημύρες και θα έχουμε και τεράστιες ε, γεωργικές εκτάσεις ε, οι οποίες ε, θα αλλάξουν. Εκεί που υπήρχαν δεν θα υπάρχουν και το ανάποδο. Θα υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι. Ε, όταν υπάρχει διοξίδιο του άνθρακα, ας πούμε, ε, μπορεί να έχουμε περισσότερα φυτά. Ε, στην παγκόσμια ιστορία φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχαν ε, κάποιες φάσεις που ήταν ε, πιο θερμό άλλες που ήταν σαν τη δική μας. Δεν ήταν και η χειρότερη εποχή λοιπόν αυτή. Επίσης, τι θα κάνει η Κομισιόν για να φέρουμε ξανά στον κύκλο το διατροφικό κάποια τρόφιμα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα, για παράδειγμα, έχουμε τις ζωοτροφές οι οποίες υπό συγκεκριμένε συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τι γίνεται με, το, ε, ζωικό, με τις ζωικές πρωτεΐνες. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν αρκετά να φάνε και το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα της παραγωγής, αλλά της αναδιανομής. Όταν έχουμε 10 εκατομμύρια τόνους ε, εκεί στις αποθήκες και δεν μπορούν να φάνε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι η Κομισιόν κάτι θα πρέπει να κάνει για την πείνα στον κόσμο και αν δούμε ποιες είναι οι προοπτικές ε, για το μέλλον, Νομίζω ότι σε αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα δεν έχουμε επαρκώς εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες. Ε, Ωραία, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ο διευθυντής Μπέλα έχει διάφορα να μας απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω. συμφωνώ και εγώ πλήρως με αυτό που είπατε για την σχέση τη παράδοση με την καινοτομία. Και αν την ξαναχρησιμοποιήσω θα σας επικαλεστώ. Υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβει υπόψη του το Κοινοβούλιο εξαιτία του θεσμικού του ρόλου. Πρώτα απ' όλα είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη επένδυση, να αυξηθεί η επένδυση σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας. αν συγκρίνουμε τις ε, επενδύσεις, τις κρατικές στην ε, έρευνα για τη γεωργία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και των ανταγωνιστών μας όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα αφετέρου είμαστε πολύ πίσω. Επομένως πρέπει να δούμε ε, πώς, πώς θα, θα φτάσει αυτή η γνώση και αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας στους αγρότες. κάποιος μέλος του Κοινοβουλίου ρώτησε τελικά σε τι είδου γεωργία θα καταλήξουμε. Θα φτάξουμε, φτιάξουμε τεράστια εργοστάσια και τεράστιες εκμεταλλεύσεις. Όχι. Αυ, αντιθέτως, αυτή η τεχνολογία θα μας επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε στην, στην τοπική οικονομία, στην τοπική μικρή εκμετάλλευση, γιατί δεν θα χρειάζεται πια να δημιουργήσει κανείς μεγάλες εκμεταλλεύσεις ή εργοστάσια. Ε, αντιθέτως, πηγαίνουμε προς μια τάση ε, μικρότερων εκμεταλλεύσεων, μικρότερων επιχειρήσεων. Ε, γιατί έχει κανείς τα τεχνικά πια εργαλεία να το κάνει. Έτσι, η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουμε τις κοινωνίες μας και τις τοπικές οικονομίες μας με όποιον τρόπο το επιθυμούμε. Και ίσως είναι η πρώτη φορά με τη βιομηχανική επανάσταση που μπορούμε να το πούμε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν, η αύξηση των επενδύσεων που χρειάζεται. Το δεύτερο, ε, και το ανέφεραν αυτό ορισμένοι βουλευτέ, είναι ότι η γνώση αυτή πρέπει να φύγει από το εργαστήριο και να φτάσει στα χέρια των γεωργών ε, η μεταφορά αυτής της έρευνας στην πράξη είναι και αυτή η παραγωγή γνώσης και αυτό σημαίνει ε, μια σειρά από πράγματα. Με ρωτήσατε για παράδειγμα αν συμμετέχουμε στην μεταρρύθμιση και στον εξυγχρονισμό της ΚΑΠ. Ναι, ε, συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους και ένα από τα ερωτήματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς αυτά τα δεδομένα, αυτές οι τεχνολογίες και αυτές οι πρακτικές που έχουμε εντοπίσει θα μπορέσουν να μεταφερθούν, να αξιοποιηθούν και μέσω των εργαλείων που μας δίνει η ΚΑΠ να φτάσουν στους γεωργούς. Ε, να χρησιμοποιήσουμε την ΚΑΠ δηλαδή έτσι ώστε να φτάσει αυτή η γνώση στους ε, γεωργούς. έτσι ώστε να, γνωρίζουν, να, χρησιμοποιούν όλα όσα μπορούμε να γνωρίζουμε για τις οδιές στην καθημερινή τους πρακτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα συνάντησα κάποιου εκπροσώπους από το Μπολιό που, ε, όπου υπάρχει μια σχολή ε, ε, γεωπόναν και διαπιστώνω ότι πολλοί από αυτούς είχαν την επιθυμία να δημιουργήσουν γεωργικές επιχειρήσεις αλλά έχουν, βρίσκονται σε δυσμενή θέση και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην ίδιο επίπεδο πληροφορίας όπως κάποιος που ζει στην πόλη χρησιμοποίησα πριν από λίγο την φράση βιοοικονομία. Ε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσιοποίησε την ε, αξιολόγηση της, μια, μια έκθεση για τη βιοοικονομία την προηγούμενη εβδομάδα και θα μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε το θέμα πιο αναλυτικά αν το επιθυμεί η Επιτροπή σας. Αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε μια σειρά εργαλείων σε μια νέα γενιά ε, γεωργών και κτηνοτρόφων ε, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν ε, αυτά τα εργαλεία για να δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο, πια στην Ήπεθρο, στις τοπικές οικονομίες να βελτιωθεί η, και, για να, η, γεωργική οικονομία και να πάει προς τον, την κατεύθυνση της βιοοικονομίας. Έχουμε μια επιλογή στα χέρια μας. Γιατί βεβαίω υπάρχουν τα ρομπότ, υπάρχουν τα drones, τα βλέπουμε αυτά, έχουμε φωτογραφίε. Το ερώτημα όμω που τίθεται είναι τελικά ποιο είναι αυτό ο οποίο παράγει προ τη θέμενη αξία. Δεν είναι ε, στην τοπική οικονομία που βρίσκεται ε, ο Γεωργό που έχει το χωράφι, που έχει το έδαφο που πρέπει να διαχειριστεί, που έχει το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το... Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι πρόκειται να γίνει μια μετα... μετάβαση, μια αλλαγή ε, ίσως ορισμένοι να ίσουν την εξή κριτική, να θεωρήσουν ότι οι ιδέες αυτές αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Όμως εγώ πιστεύω ότι στην πραγματικότητα αυτά τα εργαλεία, αυτές τις τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να πάμε πιο κοντά στους ανθρώπους της υπαίθρου, πιο κοντά ε, ε στα, στο, στους μικρούς παραγωγούς. Στην Κίνα το κράτος ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει και τι, τους παραγωγούς επειδή κατέχει το έδαφος μέχρι την πώληση των αγαθών. Επομένως το κράτος είναι εκείνο που στην Κίνα θα φροντίσει και θα επιβάλλει αυτές τις αλλαγές και θα επιβάλλει αυτές τις τεχνολογίες. Εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτό για να μην μείνουμε πίσω, να μην μείνουμε 10 χρόνια πίσω. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ λοιπόν είναι ένας τρόπος, ε, η μεταφορά τεχνογνωσίας είναι επίσης ένας τρόπος που πρέπει να αξιοποιηθεί και ε, κάτι ακόμα είναι τα δίκτυα των γεωργών, το δίκτυο Άκρη για παράδειγμα, μέσω του οποίου μπορούμε να απευθυνθούμε σε πολλούς Ευρωπαίους ε, παραγωγούς. Και άλλα προγράμματα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί να δημιουργούνται, όπως ένα εράσμος για τους γεωργούς για παράδειγμα. Κύριε αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι το έλλειμμα πρωτεϊνούχων ε, τροφίμων. Δεν ε, είμαστε εμείς ως Επιτροπή υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που δημοκρατικά λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα ή τα κράτη-μέλη. Ε, λειτουργούμε σε ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και ζούμε σε ένα συγκεκριμένο κόσμο. Ε, υπάρχουν τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες ε, προκύπτουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εμείς θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές. Για παράδειγμα, μικροάλγη ε, και οι αλλαγές που διαπιστώνουμε στον τομέα της αλίας τα τελευταία χρόνια. Πράγματα που μπορεί κανείς να κάνει όχι στις ακτογραμμές αλλά πιο στη, στην, ε, στη θάλασσα παράδειγμα ε, ενελεκτικέ ε, ε, ποικιλίε, άλλες σοδιές. Και αυτό με φέρνει στις παρατηρήσεις του κ. Φλάνακεν. και εγώ παιδί της πόλης είμαι, αλλά η οικογένειά μου είχε σχέση με τη Γεωργία στα drones Το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι περνάμε σε μια εποχή, σε έναν αιώνα, είτε μα αρέσει ή όχι, τη βιοτεχνολογία. Και θα, θα, θα, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Γίνεται ένα σημαντικό δημόσιο διάλογο για το πώ προ τα πού τελικά θέλουμε να πάμε. Και με τη ε, γεωργία και με τα τρόφιμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι διαδικασίε θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από την επεξεργασία των δεδομένων. Υπάρχει πλέον ήδη η δυνατότητα να μπορεί να συνδυάσει δεδομένα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, για παράδειγμα την ποιότητα του εδάφου, το, το, το, τα ύδατα, τον αέρα, ε, τα, δυνατότητε που έχει κάθε ποικιλία και τελικά όλα αυτά να τα συνδυάσει και να τα δώσει επεξεργασμένα σε έναν γεωργό έτσι ώστε να βοηθήσει, να, βοηθήσει να λάβει τι αποφάσει του για το πώ καλλιεργεί. Ε, όλα αυτά μπορεί κανείς να τα αξιοποιήσει για να βοηθήσει τοπικά μια τοπική παραγωγή. Ε, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάμε προς περισσότερο αυτοματισμό στην ε, ε, ε, οικονομία. Υπάρχει η επιλογή ανοιχτή μπροστά μας. Θέλουμε να έχουμε ε, γεωργούς, θέλουμε να έχουμε ύπεθρο, θέλουμε να έχουμε ε, τοπικούς παραγωγούς και φαντάζομαι ότι όλοι μας εδώ τουλάχιστον περισσότερο εδώ δίνουμε την ίδια απάντηση επόμενο ερώτημα που μετέθη είναι μήπως όλα αυτά είναι υπερβολικά high-tech υπερβολικά υψηλή τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέγγιση που έχει είναι ότι επιδιώκουμε να έχουμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μα, όλα να είναι ανοιχτά. Υπάρχουν παλαιότερε ε, τέχνικε, υπάρχουν περισσότερε παλαιότερε ποικιλίε, οι οποίε προήλθαν από τη μόνο καλλιέργεια. Ε, ίσως κάποιες από αυτές να μπορούν να βοηθήσουν στα ζητήματα της ανθεκτικότητας. Ίσως κάποιες ποικιλίε να, να έχουν προκύψει να είναι πιο ανθεκτικές. Και το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε είναι αν θα πρέπει να, αναρωτηθ, να ε, με, το, με την κλιματική αλλαγή. Νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ο πλανήτης Γη μια χαρά θα είναι. Το ερώτημα είναι οι άνθρωποι που θα ζουν πάνω του. Εάν ε, δεν γνωρίζουμε τελικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρώτος όταν σκέφτηκαν την Πολωνία και ορισμένα από αυτά που είπατε πράγματι αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, γιατί πράγματι εκεί, στην Πολωνία, στην κεντρική Ευρώπη, αυξάνεται η περίοδος του χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να καλλιεργήσουν. Αλλά ξεκινάνε αυτές οι περιοχές τώρα να έχουν πρόβλημα με τη διαχείριση των υδάτων, για παράδειγμα. Ε, οι τα νέα συστήματα ε, κυκλώνων που για πρώτη φορά είχαμε στην Ευρώπη να μας επηρεάζουν. Γιατί συνέβη αυτό. Γιατί έφτασε η θερμοκρασία του νερού στον Ατλαντικό στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και με, τους, τα ρεύματα του, ε, των ανέμων αυτό δημιουργεί κυκλώνες. Επομένως, η παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη ζεσταίνει τον νερό των ωκεανών παγκοσμίω και αυτό δημιουργεί κλιματικά φαινόμενα τέτοιου χαρακτήρα ή φωτιές δασικές στην Πορτογαλία. Επομένως, όλα αυτά συνδέονται, είναι αλληλοεξαρτώμενα, ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησης του καθενός πάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Άρα καλά θα κάνουμε να έχουμε ένα σετ εργαλείων για να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Την ε, επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει και θα ξεκινήσει μια σημαντική πρωτοβουλία για την ποιότητα των εδαφών στην Ευρώπη, για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των εδαφών, γιατί εάν κάποια, κάποια περιοχή ε, καταλήξει να έχει ποιότητα σε εδάφη, πάει. Ε, δεν υπάρχει τρόπος, είναι πολύ δύσκολο πια να επανέλθει. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε με ε, τα, τη σπατάλη των τροφίμων, τα απορρίμματα υπάρχουν μια σειρά μέτρων μέσω της ΚΑΠ και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ε, είτε ήδη από, το, από την φάρμα, από το επίπεδο του αγροκτήματος όπου βοηθούμε να χρησιμοποιούνται τα απορρίμματα για άλλους σκοπούς, ε, τα νητρικά, για τα λοιπάσματα και αντίστοιχους κανονισμούς προσπαθούμε να περάσουμε αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση ε, των επεξεργασμένων τροφίμων και για την αποφυγή χρήσης ε, υλικών τα οποία τελικά αποδείχθηκαν να μην είναι ασφαλή. Ε, εξετάζουμε επίσης με πιλωτικά προγράμματα πώ μπορεί σε δημοτικό επίπεδο, σε τοπικό ε, επίπεδο, τα αστικά απορρίμματα να μπορούν να αξιοποιούνται έτσι ώστε να μην φτάνουμε στους χιτά, να μην χρειάζεται να, ε, ούτε να τα, θάβουμε ούτε να τα καίμε αλλά να τα αξιοποιούμε ως υλικό, ω πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργεια. Και η τελευταία ερώτηση με ρωτήσατε για την Αφρική και όχι, συγγνώμη, με ρωτήσατε για το ζήτημα της αναργίας και για τη δημιουργία θέσεων εργασία στον τομέα τη γεωργία. Σε γενικές γραμμέ αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μειώνεται ο αριθμό των γεωργών. Όμως όλα αυτά βασίζονται στις προβλέψεις που μπορεί να κάνουμε αυτή τη στιγμή για, το, ε, για το ποιες θέσεις τι είδου δουλειέ υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι στα επόμενα 20-30 χρόνια τι είδου δουλειέ θα υπάρχουν στον τομέα της γεωργικής οικονομίας. Εάν, για παράδειγμα, ο τομέας της κατασκευής, των κατασκευών, ε, μεταβληθεί και αυτό και αξιοποιεί ε, βιολογικά υλικά, ε, αξιοποιεί τη δασοκομεία, ως ένα τρόπο μείωσης των εκπομπών του, ε, των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό θα δημιουργήσει ένα διαφορετικό τομέα, αν θέλετε, διαφορετικό είδο θέσεων εργασίας. με τη στρατηγική του 2012 για τη βιοοικονομία είχαμε προβλέψει μικρό αριθμό θέσεων εργασίας περίπου 700 σε αυτόν τον τομέα. Δεν, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς τον αριθμό, αλλά εάν έχουμε κάποιες προβλέψεις, αν έχουμε κάποια αριθμητικά, αριθμητικά στοιχεία θα φροντίσω να σας τα κοινοποιήσω. Και έρχομαι τώρα λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα που είχε σχέση με την Αφρική. Ε, και πάλι, εμείς που κάνουμε έρευνα και ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την καινοτομία. Δεν είμαστε αυτοί που τελικά παίρνουμε τις αποφάσεις για το πώς αυτές οι καινοτόμες λύσεις θα αξιοποιηθούν από μια τοπική κοινότητα. Ε, στην Ευρώπη έχουμε ένα δημόσιο σύστημα ε, έρευνας. Ένα ε, σύστημα έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση η οποία τελικά παράγει κάποια αποτελέσματα που θεωρούμε ότι πρέπει να φτάσουν σε αυτούς που, είναι, που έχουν τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν η σχέση μας με την Αφρική είναι διαφορετική. Εμείς ε, ε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε στη συνεργασία μας με τις αρχές των Αφρικανικών κρατών εάν υπάρχει κάποιος τομέα έρευνα ο οποίος γίνεται στην Ευρώπη και ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από αυτούς γιατί το ερώτημα που μας απασχολεί και τους μεν και τους δε είναι πώς μπορούμε να φροντίσουμε η παραγωγή τροφίμων να ανταποκριθεί στην αύξηση του πληθυσμού. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα ιδιαίτερα για την υποσαχάρια Αφρική όπου οι φυσικοί πόροι παραμένουν ίδιοι αλλά πρέπει να ε, τραφεί ακόμα ως όλο και μεγαλύτερο ε, πληθυσμό. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, John. Ευχαριστώ, Διευθυντά. Τζον Μπέλ, πολύ ε, ενδιαφέρουσα εισήγηση και η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πραγματικά και ελπίζουμε να έχουμε τέτοια σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της ε, βιομηχανίας των, των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Αντίο, Τζον, στο επανειδή. Λοιπόν, θα περάσουμε στο σημείο 12 της ημερησίας διάταξης, η απαλλαγή 2016, Γενικός Προπολογισμός της Ένωσης. Όπως ίσως θα θυμάστε από αυτό που κάνουμε και παλιό ε, τις προηγούμενες χρονιές, η Επιτροπή Γεωργίας αποφάσισε να εκπονήσει γνωμοδότηση για την απαλλαγή για το 2016. Ε, η Γεωργία ε, καταναλώνει ένα σημαντικό κομμάτι του προπολογισμού, όπως είναι γνωστό, και γι' αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Η δικιά μας εισηγήτρια στην ε, Επιτροπή για τον προπολογισμό και για την απαλλαγή θα μας δείξει, ε, θα μας παρουσιάσει μάλλον την γνωμοδότησή της. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 27 Νοεμβρίου στις 13, μία το μεσημέρι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κατά βάση αυτή η απαλλαγή έχει μια σειρά θετικών πραγμάτων που καλό θα ήταν να αναφέρουμε. Έχουμε μείωση των λαθών και παραδοσιακά βέβαια υπάρχουν περισσότερα λάθη σε σχέση με τις ε, ε, άμεσες πληρωμές, ε, στην γεωργική ανάπτυξη σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές, όμως γενικά η ανάπτυξη έχει πέσει από τα 5,3% στα 4,9%. Και εδώ να πω ότι είχαμε μιλήσει για 6% ε, λάθη στην αρχή και ευτυχώς μείναμε στο 5,3% με κάποιες ε, τεχνικές τροπολογίες διορθώθηκε αυτό. Σας ευχαριστώ για τα αυξημένα ποσοστά στην γεωργική ανάπτυξη ε, να πω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και έχουμε τονίσει στη θέση μας ξεκάθαρα ότι δεν είναι πάντα ε, το θέμα θέλησης έχει να κάνει με τις νομικές προϋποθέσεις. Να πω επίσης ότι παρόλο που είναι πειρασμός, η απαλλαγή δεν είναι ο σωστός τόπος για να μιλήσουμε για τη γενική κατεύθυνση και προσανατολισμό της γεωργικής πολιτικής. Υπάρχουν συγκεκριμένες εκθέσεις για αυτό το θέμα. Μπορούμε μέσα από εκεί να το κάνουμε. Έχουμε τους νέους γεωργούς ε, και με αυτούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της γεωργικής ε, γης και του γεωργικού τομέα στο μέλλον. Για την απαλλαγή να πω ότι και η Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο ακριβώς τα ίδια νούμερα έδωσαν για τα λάθη και παρόλο που χρησιμοποιούν άλλες ε, ε, μεθόδους και παρόλο που η Κομισιόν ε, σε περίπου 500 ελέγχους και το ελεκτικό συνέδριο 380. Γενικά ε, θα πρέπει να δούμε αναλογικά αν είναι πολλά τα χρήματα που δίνονται, δηλαδή οι έλεγχοι να μην κοστίζουν περισσότερο από όσο αξίζουν τελικά. Μετά για το greening ε, υπάρχει ε, αρνητική επίπτωση στο ποσοστό λαθών, όμως είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Για το θέμα του περιβάλλοντος βλέπουμε μία βελτίωση η οποία μόνο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορεί να παρατηρηθεί και να αξιολογηθεί. Γενικά βλέπουμε ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Είναι η επόμενη εβδομάδα. Ε, η προθεσμία μας. 24 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, οπότε θα ζητήσω από τους συναδέλφους να μου πούν τι υποστηρίζουν και τι δεν υποστηρίζουν. Θα το ακούσουμε σύντομα και με τις παρεμβάσεις τους. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες ε, πληροφορίες και αυτό έχει μειώσει πολύ το ποσοστό των λαθών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση γενικά είναι θετική και να σας πω ότι τα υψηλά ποσοστά λαθών δεν έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπήρχε αμέλεια ή κακοδιαχείριση των ε, ε, χρημάτων των ε, φορολογουμένων, Απλώς ε, είναι τεχνικά τα ζητήματα, δηλαδή κάποια χρήματα μπήκαν σε λάθος προϋπολογισμό ή έγιναν κάποιες ε, αναβολές, ε, δεν έγινε σωστή αξιολόγηση λογαριασμών, δεν ήταν κάποια εγκληματική δράση δηλαδή, υποδήγησε σε όλα αυτά. και όταν έγινε η εγιναν καποιες αναβολες δεν εγινε σωστη αξιολογηση λογαριασμων δεν ηταν καποια εγκληματικη δραση δηλαδη υποδηγησε ολα αυτα και οταν εγινε η διορθωση Γενικά μπορέσαμε, όταν κάναμε τον απολογισμό και ξεκαθαρίσαμε τους λογαριασμούς, μπορέσαμε να λύσουμε αυτά τα λάθη. Γιατί θα ήταν ε, λάθος ε, να λέγαμε ότι αυτά τα νούμερα είναι συνώνυμο απάτης ή κάποιας ε, διεφθαρμένης στάσης από την πλευρά των αρχών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ε, εισηγήτρια την κυρία Κάντεμπαχ. Όντως έκανε μια παρουσίαση γρήγορα και πολύ συγκεντρωμένα, να την ε, συγχαρώ. Ήταν πολύ καλό, προς τους φιλικό προς τους βουλευτές αυτό, δεν χρειάστηκε καν να το διαβάσουμε, ήταν πιο εύκολο να το ακούσουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία Κανείς θα μπορούσε να σχολιάσει. Και εγώ ο ίδιος μπορώ να πω ότι υπάρχουν αυτά τα ποσοστά λαθών στην γεωργία, μεν, αλλά τα ποσοστά είναι σχεδόν μηδενικά. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο greening, ε, να γίνει πιο οικολογική δηλαδή η γεωργία. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να συγχαρούμε κυρίως τους γεωργούς οι οποίοι πρέπει να παλέψουν με την ε, ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και τα καταφέρνουν. Βλέπουμε ότι μειώθηκε εκτάσεις, τα λάθη στις γεωργικές εκτάσεις. Ε, η δική μου θεωρία είναι ότι συνήθως τα προγράμματα για αυτά τα θέματα είναι πολύ περίπλοκα και δεν πάνε στην σωστή πελατεία. Αν αυτό γινόταν σε αιτήσια βάση, αν έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί κάθε χρόνο να παλεύουν με την γραφειοκρατία, ε, υπάρχει ένα ποσοστό προσαρμογής που πρέπει να γίνει ε, Άρα αν μειώσουμε την γραφειοκρατία θα έχουμε καλύτερα ε, αποτελέσματα. Είναι αυτό έκκλησή μου προς αυτούς που κάνουν τα προγράμματα, να τα κάνουν πιο φιλικά προς το χρήστη. Επίσης, να πω ότι τα περισσότερα λάθη που έχουμε εδώ δεν είναι διασπάθηση δημόσιου χρήματος ή διαφθορά. Το λέω και εγώ υπόθηκε ήδη. Να πω και πάλι, συγχαίροντας την κυρία Κάντεμπαχ, ότι ήταν πολύ καλό είναι πολύ καλό το κείμενο της θέσης, μπορεί κανείς να το καταλάβει, να το διαβάσει, να το πάρει σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ και τώρα συνάδελφος Μπέλτερ, σκιώδης επίσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Κάντενμπαχ ε, για τα ε, γνωμοδότησή της. Το ποσοστό σφάλματος έχει εκ νέου μειωθεί. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Και όπως είπε ο κύριος Γιάρ, είναι ένα επίδευμα των γεργών και των μηχανισμών ε, καταβολής των ποσών Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία. Μπορούμε να προσθέσουμε κάτι σε σχέση με τα θετικά στοιχεία, για παράδειγμα διορθωτική δυνατότητα, corrective capacity, για κινδύνους δηλαδή που μπορεί ακόμα περισσότερο να μειωθούν ε, και μπορούμε επίσης να αναφερθούμε στην βελτίωση του συστήματος ε, εντοπισμού, του LPS, είναι πιο συγκεκριμένο και επιτρέπει τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Χαίρομαι ήδη λοιπόν για τη συνεργασία την Καρποφόρα και ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Και εγώ ξεκινώ ευχαριστώντας την εισηγήτρια για το σχέδιο χρωμοδότησής της, το οποίο είναι πολύ ισορροπημένο. Ε, νομίζω πως η κατεύθυνση στην οποία ε, οδηγεί είναι πολύ θετική. Το ποσοστό σφάλματος στις πληρωμές στο πλαίσιο της γερικής πολιτικής έχει μειωθεί ε, σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα, είναι πολύ θετικό. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας ρωτήσω, να μου επιτρέψετε να θέσω μια άλλη ιδέα επιπλέον των όσων μας είπε η συγγετρία. Θα μπορούσαμε κάποια σημεία ίσως από αυτά να τα προσθέσουμε. Για παράδειγμα, η Κομισιόν θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα σύστημα ελέγχων που θα επιτρέπει τη μείωση του διοικητικού φόρτου βλέπουμε ότι ο Γιώργος υποχρεούται να προβεί σε διάφορους ελέγχους, σε διάφορα επίπεδα. Κατά τη γνώμη μας αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί επιπλέον ε, για την αναθεώρηση των ελέγχων. Σε αυτή την αναθεώρηση δεν θα μπορούσε να γίνει η βάρος της, της, ε, ε, του δίκαιου χαρακτήρα των ελέγχων Έλεγχος βασισμένος στους κινδύνους πιστεύω πως είναι ένα ε, σημαντικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε κάποια πλαίσια στο περιθώριο σφάλματος, ενώ πολλά σφάλματα οφείλονται στον περίπλοκο χαρακτήρα ε, ωστόσο παραμένει σφάλμα και καταγράφεται ως σφάλμα. Και κάποιος διακινδυνεύει την επιβολή κυρώσεων. Εδώ θα πρέπει να εισάγουμε κάποια ευελιξία και αναλογικότητα που δεν επικρατεί πάντοτε. Πάντως ευχαριστώ την εισηγήτρια ακόμη μια φορά γιατί η πρότασή της είναι πολύ ισορροπημένη. Ίσως λοιπόν λίγο μεγαλύτερη προσοχή να δώσουμε στο Grazie. μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου. Ευχαριστούμε κύριε Τάκουλα και τώρα ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εξαιρετική ε, η γνωμοδότησή σας. Ε, αντίθετα από τον ε, κύριο Μπέλντερ, εγώ θα έλεγα ότι το 3 όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει εδώ, αλλά αν μπορείτε να το βάλετε και να το υπογραμμίσετε για να το τονίσετε ακόμη περισσότερο να το κάνετε, γιατί είναι μια εντοπιστική κατάσταση όπου βλέπουμε ότι έχουμε καταλήξει σε μια κατάσταση όπως αυτή που δηλώνεται εδώ στο 3 ε, στο σημείο 3. Για τα άλλα σημεία 1, 2, 4 και 5 λένε ότι το λάθος είναι Ε, είμαστε λίγο άνθρωποι λοιπόν, θα κάνουμε σφάλματα. Ε, δεν είναι πάντοτε η θελημένα, αλλά ένα από τα πράγματα που προκαλούν τα σφάλματα είναι η περιπλοκότητα των συστημάτων και μία ρήξη στην αλυσίδα επικοινωνία ανάμεσα στην Επιτροπή, τι εθνικέ κυβερνήσει και τον Γεωργό. Γιατί έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσει όπου οι κανόνες και οι κανονισμοί ήρθαν, ε, δόθηκαν συγκεκριμένα δελτία στα Υπουργεία το... Γεωργίας των χωρών μας και μετά αυτό που δόθηκε στα Υπουργεία δεν ήταν το ίδιο που δόθηκε και στους Γεωργούς. Επίσης, σε άλλη περίπτωση, κάποιος έλεγε ότι του έβαλαν πρόστιμα επειδή το σύστημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Του ζήτησαν να πάει σε κάποιο σύμβουλο. Και η απάντηση ήταν ότι εγώ ίδιος ήμουν σύμβουλος μέχρι πριν από λίγους μήνες και ούτε εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Κοιτάξτε, όσο πιο περίπλοκο είναι το σύστημα, τόσο περισσότερα θα σφάλματα θα κάνουν οι άνθρωποι και ε, τη μόνη λύση είναι η απλοποίηση. Ευχαριστώ. Ο Μισελ Νταντάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συγγήτρια για την γνωμοδότησή της και επανέρχομαι σε μια φράση που χρησιμοποίησε και που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική διότι ακούμε πολλά για το πρασίνισμα. Η συγγήτρια μας είπε όμως πως ήταν ακόμα πολύ νωρίς, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μετρήσουμε τις απτές ε, συνέπειες επί τόπου και τον αντίκτυπο στη βιοπικιλότητα και αυτή ε, η σκέψη θα πρέπει να υπάρχει και στην έκθεση. Όπως επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτό που έχουμε ήδη την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, ε, ε, συγγνώμη, τον πρόεδρο το συνεδρίου, το γεγονός δηλαδή ότι οι αναλύσεις του συνεδρίου αφορούν το τελευταίο λεπτό του ευρώ, πού χρησιμοποιήθηκε, αλλά όχι αν ήταν σωστή αυτή η χρήση. Δεν ελέγχεται η σωστή χρήση. Ε, αν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, θα μας βοηθήσει να είμαστε λιγότερο ανόητοι σε ορισμένους από τους ελέγχους που γίνονται επί τόπου. Ευχαριστώ, ο Άλμπερτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τη συνάδελφο Κάντεμπαχ για την πολύ καλή έκθεση. Να συμφωνήσω και με τους ε, συναδέλφους ότι θα υποστηρίξω πλήρως αυτή την έκθεση. Κυρία Κάντεμπαχ, ε, θα ήθελα να πω σε σχέση με την έκθεση ότι όταν μιλάμε για λάθη, και το είπαν και οι συνάδελφοι, ε, έχουμε ε, μια διαφοροποίηση. Αυτά που έχουν επιπτώσεις ε, στους φορολογούμενους και αυτά που έχουν μια άλλη αξιολόγηση. Φαίνεται ότι κάποιοι ξέχασαν να γράψουν κάποιες βάσεις δεδομένων και αυτό ε, του στήχησε κά, κάποια πράγματα, όμως ε, κάποιες ε, σε αυτή την περίπτωση οι φορολογούμενοι γλίτωσαν χρήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό θα είναι να έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία αυτές τις δύο κατηγορίες. Επιπτώσεις που έχουν η μία κατηγορία είναι τα λάθη που έχουν επιπτώσει στους φορολογούμενους και η άλλη αυτά που δεν έχουν καμία τέτοια επίπτωση. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε ένα σύστημα τόσο περίπλεκο, όλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ ένας γεωργός, ας πούμε, δεν κατέθεσε σωστά στις βάσεις δεδομένων και τελικά τιμωρήθηκε. Όταν κάποιος πάει το παιδί στο σχολείο και ξεπερνά το όριο ταχύτητας, παίρνει ε, κλίση. Ε, και εδώ στη Γεωργία ε, το ίδιο πρέπει να γίνεται και πρέπει εντατικά να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Bene, grazie colleghi, sono intervenuti tutti. Adesso darei la parola alla Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πήρατε όλοι το λόγο. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ε, εκπρόσωπο της DG Agri, κυρία Πόρτσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς για όλα τα θετικά σχόλια, για όσα ε, ακούσαμε φέτος, ε, να πω ότι όλο το ποσοστό λαθών ήταν 2,5% είναι το ίδιο που είχε και η DG Agri ε, πριν από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Άρα φτάσαμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αντί να μιλάμε για ποσοστά λαθών, να μιλάμε ότι έχουμε αξιοπιστία για περισσότερο από το 97,5% των δαπανών. Και κάπου εκεί να τελειώνει. Ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότηση. Τώρα για τα διάφορα που είπατε δεν θα κάνω και πάρα πολλά σχόλια. Μπορεί να ξέρετε ότι ο Επίτροπος Χόμπαγκαν θα πάει την επόμενη Τρίτη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για να συζητήσει όλα τα θέματα που θέσατε μεταξύ αυτών και την κατανομή των άμεσων πληρωμών. Όπως είπατε και πολλοί από εσά βέβαια, ε, το ποσοστό λαθών δεν δείχνει ότι υπάρχει απάτη στον ε, της Γεωργίας. Αν δείτε την τελευταία έκθεση Όλαφ που εξετάζει το ποσοστό της απάτης είναι ε, το χαμηλότερο ποσοστό σε οποιοδήποτε σημείο του προϋπολογισμού. Άρα τα νούμερα πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Μιλάμε για σφάλματα, ε, συστήματα ελέγχου που δεν λειτουργούν σωστά, αλλά όπως και να έχει και για την DG Agri με το 1,7% στον πρώτο πυλώνα από το ελεκτικό συνέδριο είναι πολύ καλά τα νούμερα. Να πω ότι συνολικά το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά από το 1994 έκανε μία ε, ε, γνωμοδότηση ε, αυτού του είδους για, για την ε, γεωργία. Στο παρελθόν ήταν πάντοτε αρνητική η έκθεση. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη γνωμοδότηση εδώ και θα υπάρξει και περισσότερη συζήτηση από τον Επίτροπο, με τον Επίτροπο Χόγκαν την επόμενη εβδομάδα. αλλά... Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα σχόλια. Και τώρα θα δώσω στην Κάρεν και πάλι το λόγο. Ναι, να ευχαριστήσω για τις σκέψεις ε, των συναδέλφων. Θα συμπληρώσω τα, όλα, τα όσα έχω κάνει με αυτά που μόλις μου είπατε και ευχαριστώ και για την ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο Χόγκαν. Ευχαριστούμε την Κάριν. 27 Νοεμβρίου προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών ε, στη μία το μεσημέρι. Και τώρα περνάμε στο πρώτο τελευταίο σημείο, το 11 της ημερησίας διάταξης. Το επόμενο έχουμε παρουσίαση από προ, εκπρόσωπο της Κομισιόν όσον αφορά την παράταση της διάρκειας των δικαιωμάτων των παραγωγών σπαραγγιών, βολβών και λοιπόν βολβών ανθέων. Συζήτηση λοιπόν που θα κάνουμε σήμερα και δίνω αμέσως το λόγο στην Άννη που θα μας παρουσιάσει αυτό το θέμα και μετά θα ακούσουμε την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και τις παρατηρήσεις της. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de Europese Commissie heeft tot nu toe geen actie ondernomen om het kwekersrecht voor bloembollen, asperges en houtachtige struiken. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσω την, ε, το αίτημα που μας υποβλήθηκε για να ε, ε, αυξηθεί η περίοδος προστασίας για αυτές τις ποικιλίε φυτικών ποικιλιών για τους βολβούς, άνθεων, χαμόδεντρα και παρά το γεγονό ότι, ότι ε, μάλλον αυτή τη στιγμή που πλήθηκε αυτό το αίτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει, θα πρέπει να δει ε, πώς θα αντιδράσει σε αυτό. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματα των ε, βελτιωτών αλλά να φροντίσουμε των, των, των ποικιλιών δηλαδή, αλλά να φροντίσουμε ταυτόχρονα και την προστασία των γεωργών. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο ε, Ολλανδικού ενδιαφέροντος παρά το γεγονό ότι το αίτημα έχει υποβληθεί από, στην Ολλανδία. Αλλά έχουμε και καλλιέργειες ε, φράουλας στην Πολωνία οι οποίες θα επηρεαστούν από οποιαδήποτε απόφαση, τα μύρτιλα στην Ιταλία. Επομένως, συζητούμε το ζήτημα αυτό με βάση την νομοθεσία και συγκεκριμένα τον κανονισμό 194 ε, του 2000, στο άρθρο 19, παραγραφούς 1 και 2. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ε, παραγωγούς και προτείνουμε την παράταση, να δοθεί παράταση σε αυτό το δικαίωμα προστασίας. Σα ευχαριστώ. Να καλωσορίσω την εκπρόσωπο της δική Santa, την κυρία Δωροθέα Αντρέ, που ήρθε ήδη εδώ επάνω. Καλωσορίσατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καλημέρα σε όλους και όλες. Ε, ευχαριστώ που μας καλέσατε για να σας εξηγήσουμε πού βρίσκεται η Κομισιόν σε αυτό το αίτημα, στο πλαίσιο αυτού του αιτήματο παράτασης της διάρκειας της προστασίας των ποικιλιών.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 Donc, il y Έχει ήδη υποβληθεί αίτημα για παράταση το 2008. Έγινε υπευλήθη το αίτημα στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ε, του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και αφορούσε τα σπαράγγια και άλλα είδη και συγκεκριμένα τις φράουλες. Το 2009 συστήσαμε μια ομάδα εργασία για να εξετάσει το θέμα με την, το κοινοτικό γραφείο, την Κομισιόν και τις οργανώσεις των βελτιωτών και καταλήξαμε ότι ήταν δύσκολο να ορίσουμε τους λόγους για του οποίους ορισμένα ήδη χρειάζονταν μια διάρκεια προστασίας μακρύτερη και ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίε από τους βελτιωτέ για να αιτιολογήσουν το αίτημα παράταση της διάρκεια προστασίας. Εν τω μεταξύ η Κομισιόν ξεκίνησε μια αξιολόγηση εξωτερική τη νομοθεσία. για, που, που κάλυψε έτη 1995 μέχρι 2011 και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινοτικού Γραφείου Βετικών Ποικιλιών ε, αποφάσισε να αναστείλει τη διάρκεια του αιτήματο. Η εξωτερική αυτή αξιολόγηση εξέτασε τη διάρκεια της προστασίας και ε, έδειξε ότι το ισχύον σύστημα λειτουργούσε σωστά, ότι η διάρκεια προστασίας μάλιστα προεκύπτει από αυτή την αξιολόγηση, ήταν ανάλογη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συστήματος, ότι ήταν συγκρίσιμη με τα εθνικά συστήματα προστασίας ότι οι βελτιωτές ζητούσαν την αύξηση της διάρκειας, αλλά αντίθετα άλλοι φορείς πίστευαν ότι η διάρκεια ήταν επαρκής. Μετά από αυτή την αξιολόγηση, μία ομάδα πυρογνωμόνων ε, ενέκυψε στα απορίσματα. Ε, αποτελείται από την Κομισιόν, τους βελτιωτές, ε, το γραφείο, γραφείο των φυτικών ποικιλιών και έγινε μια σειρά από συνεδριάσεις ανάμεσα στο 2012 και το 2015 και πρέπει να πω ότι αυτή η υπόθεση της προστασίας δεν ε, φύγει στο ομάδα εργασία των υπηρογνωμών. Ωστόσο, το 2016 έγινε επίσημο αίτημα προαράταση τη διάρκεια και υπευλήθη ε, από τον πρόεδρο του Κοινοτικού Γραφείου Φετικών Ποικιλιών προ την Κομισιόν αφορά του, τα σπαράγγια, ε, τα φράουλα, τα σμέουρα και τα μύρτιλα, όπως μας είπε και η κυρία ε, βουλευτής και τα, τους βόλβους ανθέων. Εξετάσαμε αυτήν, την, το αίτημα. Ο Γενικός Διευθυντής αναγνωρίζει φυσικά τη σημασία του αιτήματο και τη σημασία της ε, απόσβεσης ε, των επενδύσεων. Θύμισε ότι στη διάρκεια της αξιολόγησης νομοθεσίας τις θέσεις ήταν ε, μοιρασμένε ανάλογα με το ποιο έπαιρνε το λόγο και ότι άρα βεβαίω οι βελτιωτές ζητούσαν παράταση αλλά δεν το ζητούσαν όλοι και ότι θα έπρεπε να μπορέσουμε να προβούμε σε μια εις βάθος ανάλυση του αντικτύπου μιας παράτασης της διάρκειας. Όχι μόνο αντίκτυπο για τον ίδιο τον τομέα των βελτιωτών, αλλά και για ε, τους διδροκόμους και τους καταναλωτές. Αυτό που είπαμε λοιπόν είναι ότι αν ε, τροποποιήσουμε την νομοθεσία, πρόκειται για τροποποίηση του άρθρου της οδηγίας της βασικής του Συμβουλίου, αυτό έχει μπει στη Λισαβόνα και άρα θα είναι ένα αίτημα του ε, Συμβουλίου και θα είναι δηλαδή έτοιμα τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Άρα σε έχουμε συναπόφαση και ότι ε, θα είχε ανάγκη η Κομισιόν από μια σειρά από στοιχεία. Τα βλέπετε εδώ, έχετε μια ολόκληρη σειρά από στοιχεία για τον αριθμό των ποικιλιών, τη μέση διάρκεια προστασία, ε, μετά από πόσο χρόνο ε, οι ποικιλίε δεν προστατεύονται πια, ποιο είναι από πίσω, ποιοι είναι οι βελτιωτέ κτλ. Ίσως θα ήταν καλό να θυμίσουμε ποια είναι, τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Εμείς με την κοινοτική μας νομοθεσία επιτρέπουμε την διάρκεια της βελτίωσης για ε, προστασία για 20 χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις για 25 χρόνια. Οι διεθνείς συμβάσεις Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτικών ε, ε, Ποικιλιών είναι μικρότερης διάρκειας. Η μέση διάρκεια προστασίας για τις περισσότερα είδη είναι 20 ετία διεθνώς, ενώ εμείς προτείνουμε 25 χρόνια και η πιο μακρά περίοδος προστασίας σε επίπεδο της Διεθνούς Σύμβασης είναι 25 χρόνια για τα δέντρα και τα μπέλια ενώ εμείς προτείνουμε τα 30 χρόνια. Το σύστημά μας προστατεύει λοιπόν για μεγαλύτερη διάρκεια. fait hier la, euh, une euh, réponse à notre εδώ έρχεται ένα άλλο ερώτημα και λάβαμε την απάντηση του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών που μας απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και τα στοιχεία που είχαμε ζητήσει. Άρα λοιπόν από τη δική μας πλευρά δεν μπορώ σήμερα να σας πω βέβαια το τι έκανε αυτό το αίτημα γιατί μας έφτασε μόλις εχθές το απόγευμα. Βεβαίως θα το εξετάσουμε εις βάθος και αν θέλουμε να συνεχίσουμε, να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την, ε, το αίτημα παράτασης, ξέρετε πολύ καλά, όπως και εγώ, ποια είναι η διαδικασία, η νομοθετική. Πριν να στείλουμε πρόταση της Κομισιόν για τροποποίηση ενός κανονισμού Χρειάζεται μια εκτίμηση, μια μελέτη αντικτύπου. Όλα αυτά παίρνουν χρόνο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έρθουν σε διαβούλευση, όχι μόνο οι βελτιωτές, αλλά καθένας που ε, επηρεάζεται, οι καλλιεργητές, οι καταναλώτες, όλοι θα συμμετέχουν σε διαβούλευση. Όλα αυτά απαιτούν λοιπόν εις βάθος μελέτη και πολλά χρόνια πολλά κράτη έχουν ε, προτείνει ε, στο Συμβούλιο παράταση. Θα αναλύσουμε λοιπόν εάν έχουμε αρκετά στοιχεία στη διαθέσή μας ώστε να μπορέσουμε να αντισταθούμε στο Impact Assessment Board που ζητά εξονυχιστική εξέταση κάθε πρότασης και του οικονομικού και κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου για κάθε νέο αίτημα. Σήμερα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε λοιπόν ευρύτερα το θέμα γιατί μόλις το λάβαμε και θα είμαστε σε θέση να πούμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες, αλλά όχι άμεσα, γιατί πρέπει τώρα να μελετήσουμε τα πολλά και διάφορα παραρτήματα που μας ε, έχουν ε, δοθεί. Αυτή είναι η επόμενη φάση, ε, αλλά βεβαίως το θέμα αυτό θα εξεταθεί στη όπως δει και γνωρίζουμε και ε, θα, με τη δέουσα προσοχή. Λοιπόν, ευχαριστώ Πρόεδρε, μας δώσετε το λόγο. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, κυρία Διευθύντρια και τώρα θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Μπέλντερ πρώτα και μετά τον κύριο Αγγνιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε το δικαίωμα ε, του βελτιωτή είναι πολύ καλό σύστημα διότι προσφέρει μέτρα προστασίας για τις διάφορες ποικιλίε που όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν νέες ποικιλίε. Για τους βαλβούς ανθέων και για τα σπαράγγια και τα τους βολβούς ε, α, και για τα χαμόδεντρα. Ε, έχουμε πρόβλημα. Ε, μία παράταση 5 ετών θα ήταν επιθυμητή. Πιστεύω πως υπάρχει υποστήριξη από πλευρά των εμπειρογνωμόνων των εθνικών αλλά και από το Κοινοτικό Γραφείο φοιτικών Ποικιλιών με άλλους συναδέλφους εδώ θα θέλαμε η Επιτροπή να δώσει ένα θετικό μήνυμα υπέρ αυτών των αλλαγών και αυτό όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ο Στιούαρτ Αγνίου. Ευχαριστώ. Μιλάμε για την αρχή των δικαιωμάτων και της προστασίας φυτών και δέντρων είναι η μόνη πηγή εισοδήματος και υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποτυχίας γιατί μπορεί να έχουν 100 ποικιλίε ε, στην παραγωγή, αλλά αργά ή γρήγορα μπορεί από τις περισσότερες από αυτές να χρειαστεί να τις εγκαταλείψουν ε, γιατί δεν ε, είναι βιώσιμες. Αλλά τυχαία μπορεί κάποια στιγμή να πιάσουν το jackpot και το ένα. Αυτό πρέπει να καλύψει το κόστος όλων των προηγούμενων αποτυχιών. Πράγμα το οποίο δεν εκτιμάται, δεν λαμβάνεται υπόψη. Πολλές εταιρείε που το κάνουν αυτό δεν είναι κάτι τεράστιες πολυεθνικές. Ορισμένες είναι απλώς οικογενειακές επιχειρήσεις και πιστεύω πως έχουν κάθε δικαίωμα να να ζητούν κάποια αποζημίωση για την πνευματική τους ιδιοκτησία. Διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο και όλοι θα βγουν χαμένοι. Επίσης θα μπορούσαν να έχουν ε, κάτι πολύ καλό ως να το πάνε μετά στην αγορά και μετά να, αναγνω... να καλύψουν πως ένας ανταγωνιστής έχει κάνει κάτι που είναι λίγο ελάχιστα καλύτερο. Όχι τελείως καλύτερο, αλλά ένα μικροσκοπικό ποσοστό και όλοι θέλουν αυτό το ανταγωνιστή και κανείς δεν θέλει αυτό που έφτιαξαν οι ίδιοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτοί που αγοράζουν αυτούς τους πόρους, ε, ε, θάμνους και τα κτλ. αναμένουν να κερδίσουν. Γιατί λοιπόν να κερδίσουν δεν τους αρέσει να δίνουν και ένα κομμάτι σε αυτούς που το φτιάξαν, εν πάση περιπτώσει. Πριν από λίγους μήνες ε, είχα ε, είδα κοντά στο σπίτι μου ένα χωράφι με ζαγαρότεφλα που φαινόταν ε, καημένο, έτσι, καχυκτικό. Γιατί δεν κατάλαβα γιατί λέει αυτή η γη ε, δεν ήταν έφορη για αυτό το είδος της καλλιέργειας. Αν το ήξερα πριν από 40-50 χρόνια δεν θα είχα ποτέ φυτέψει εκεί ζαχαρότεφλα. Ε, ρώτησα αν είναι ανθεκτική αυτή η ποικιλία. Απλά, γιατί κάποιος είχε, ε, είχε προνοήσει για να φτιάξει μια ποικιλία που θα άντεχε σε αυτό ένα, ειδικό, ένα συγκεκριμένο σαράκι του ζαχαρότεφλου. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν, ε, ζουν παιδί. Δεν μπορούμε οι Γεωργοί να φτιάξουμε τα δικά μας τρακτέρ, δεν μπορούμε να φτιάξουμε συνθετικά ζυζανιοκτώνα κτλ. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλλιεργούμε σπόρους. Και τίποτα δεν θα σταματήσει ένα Γεωργό από το να επιμείνει σε μια ποικιλία που δεν έχει ε, ποσοστά, δεν έχει προστασία, και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν και να παραχρεώνουν ούτω ή άλλω να υπερβάλλουν, γιατί ένα γεωργό πάντα έχει την ε, επιλογή να επανέλθει και να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία για την οποία δεν χρειάζεται να καταβάλει το ποσοστό της προστασίας. Ευχαριστώ, Στιουαρτ. Τελευταία παρέμβαση, Γιουτέμα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσει. Η συζήτηση είναι ιδιαίτερα τεχνική. Ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα όμως. Νομίζω ότι υπάρχει ε, ενδιαφέρον για την ε, παράταση των πέντε ετών. Γιατί, Γιατί είναι σημαντικό να φτάσουμε σε μία ε, καλλιέργεια με αυξημένη ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένες ασθένειες. Για κάποιες καλλιέργειες αυτό ε, σημαίνει ότι θα χρειαστεί χρόνος. Δεύτερον, οι μικροί γεωργοί θα μπορούσαν να έχουν μια μεγαλύτερη προστασία και να έχουν και ωφέλη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις αυτό που θα ήθελα θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι γρήγορα ξεκάθαρη για αυτό το θέμα. Να μας πει γρήγορα αν γίνεται ή όχι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις που περιμένουν τις απαντήσεις να λάβουν υπόψη τους ε, την απάντηση. Ευχαριστούμε τον Γιάννη. Δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω το λόγο σε εσά ή πάλι στην DG Sante. Συνάδελφε Άννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή για την απάντηση που μας έδωσε. Θεωρώ όμως ότι στην Ευρώπη δεν πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε αενάως για τη Μονσάντο και όλα αυτά. Μας είπατε ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα γιατί πραγματικά έχουμε κάνει άπειρες διαβουλεύσεις ε, με τις μη κυβερνητικέ ε, και πρέπει πριν το καλοκαίρι να έχουμε ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Θα υπάρχουν επιπτώσεις ε, από αυτό το άρθρο 2. θα πρέπει να το δείξουμε αυτό. Εν μέρη με ικανοποιεί η απάντησή σας, από την άλλη όμως δεν πρέπει να σπαταλάμε και το χρόνο μας. Πρέπει να είμαστε γρήγορα πιο βέβαιοι ως Ευρώπη. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Τελευταία η διευθυντριά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αγαπητοί Ευρωβουλευτές, καταρχάς για την υποστήριξη για το γεγονός ότι θεωρείται πως είναι ευνοϊκά τα δικαιώματα ε, των κατόχων. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πίσω. Έχουμε το θέμα και θα το εξετάσουμε με βάση αυτά τα στοιχεία. Επί της ουσίας είναι ε, αυτές οι διαδικασίες βέβαια πολύ επαχθείς θα έλεγα, ε, πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να αντισταθούμε στο Pack Assessment Board για να δείξουμε ότι υπάρχει ένα θετικό συμφέρον για ολόκληρη την αλυσίδα και όχι μόνο για την αρχή της αλυσίδας ε, για να υπάρχει ε, επίπτωση όχι μόνο στους γεωργούς αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, που, αυτούς που έχουν τα δικαιώματα της παραγωγής φυτικής ποικιλία και στους καταναλωτές. Η επέκταση είναι απαραίτητη και δικαιολογημένη. Η Κομισιόν λοιπόν αν θεωρεί ότι, είναι, ότι νομιμοποιείται να υπάρχει αυτή η επέκταση θα κάνει την πρόταση σχετικά την οποία θα στηρίξει με επαρκή στοιχεία, φαντάζομαι. Υπάρχει κάποιος καιρός, ε, κάποιο μεγάλο διάστημα που έχει περάσει, γιατί πραγματικά δεν είναι τόσο απλό το θέμα, από ό,τι φαίνεται. Ε, ε για να συζητάμε από το 2008 μάλλον δεν είναι προφανές το ζήτημα. Υπάρχουν και νέα στοιχεία που προστέθηκαν, θα τα εξετάσουμε σοβαρά. Δεσμευόμαστε απέναντί σας να μπορέσουμε πριν το καλοκαίρι να σας δώσουμε στοιχεία σχετικά με το πού βρισκόμαστε για αυτό το θέμα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα... Πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχει να κάνει με την παρουσίαση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παραγωγών Τυριού και των γαλακτοκομικών ε, προϊόντων. Δεν έχουν ακόμα καταφτάσει οι ειδικοί μα σε πέντε λεπτά διάλειμμα, γιατί πρέπει να περιμένουμε τους ειδικούς.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

Bene, colleghi, allora andiamo per l'ultimo punto. Ωραία συνάδελφοι, πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησία μας διάταξης που αφορά την παρουσίαση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παραγωγών ε, ε, Τυριών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, την ΦΑΤΣΕ. Μπορείτε να ακούσετε μετάφραση και είναι καλύτερα να σβήσετε και το τηλέφωνο σας, ε, λέει ο Πρόεδρος στον ομιλητή πρόσφατη γνωμοδότηση για τον ε, προπολογισμό και η, Κομισιό, η Επιτροπή μας αποφάσισε να κάνει μια εξπόστα αξιολόγηση των πιλωτικών προγραμμάτων για να επαληθεύσει αν επενδύθηκαν σωστά οι ε, πόροι του project ε, αυτού και γι' αυτό και οι συντονιστέ αποφάσισαν να βάλουν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι ίδιοι οι του πιλωτικού προγράμματο μας ζητήσαν αυτή την ευκαιρία ε, υπογραμμίζοντα ότι ε, συνεργάστηκαν στενά με την DG Santa για να επεξεργαστούν τι καλέ πρακτικέ προς τους παραγωγούς που θα απευθύνουν στους παραγωγούς ε, γαλακτοκομικών προϊόντων μικρών διαστάσεων να εξετάσουμε την προσθέμενη αξία ε, για τις πολλέ μικρομεσαίες εταιρείε που εργάζονται στον τομέα αυτό. Ε, αυτό το τμήμα θα βοηθήσει δε, τα μέλη μας να εμβαθύνουν στις δυναμικές ε, παρουσίασης και να μας επιτρέψει να δούμε πώς τέτοιες ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε κάτι που η Κομισιόν όχι μόνο θα δεχτεί αλλά θα αποφασίσει και να τα αναπτύξει. Μετά από αυτή την παρουσίαση θα ακολουθήσει μια εκδήλωση. Non qui in Parlamento. Όχι εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά στο κτίριο Γιάννη, στον τρίτο όροφο, όπου θα περάσουμε σε, ε, ε, ε, για να δοκιμάσουμε την παραγωγή τυριών. Θα είναι και νόστιμη λοιπόν αυτή η παρουσίαση. Ε, πριν να δώσω το λόγο στον φίλο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παραγωγών Τυριού και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, να χαιρετήσω την Περνοντέ Τελάνς που είναι εδώ μαζί μας και είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Τυριού και πρόεδρος διεθνώ, της παγκόσμιας δηλαδή Συνομοσπονδίας Παραγωγών Τυριών. Α, των διανομέων, όχι των παραγωγών. Μάλιστα. Μπερνατέ, Τελάνζ. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο για την παρουσίαση του πιλωτικού προγράμματος. Έχεις το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Φρεντερίκ Μπλανσάρ. Είμαι παραγωγός ε, κατσικίσιου τυριού στην περιοχή Αλπ που είναι 30 χιλιόμετρα από τη Λιόν και φτιάχνουμε χειροποίητο τυρί εδώ και 25 χρόνια. Εδώ και 8 χρόνια ασχολούμαι με ένα δίκτυο ε, γαλακτοπαραγωγών ε, και τυροκόμων, το οποίο δημιουργήθηκε επισήμως το 2013 παρόλο που υπήρχε από το 2009. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία που είχαμε μέσω αυτού του δικτύου και χάρη στην υποστήριξη της DG ε, Santa και της Επιτροπής Γεωργίας ήταν ο Ευρωπαϊκός ε, κατάλογος, ε, οδηγός ε, για την ε, παραγωγή του τυριού και τυριού βιοτεχνικού. Μικρής κλίμακας δηλαδή, παραγωγής από παραγωγούς. Αυτό το δίκτυο λοιπόν τι εκπροσωπεί. Αυτός είναι ο χάρτης του δικτύου FACE. Έχουμε 15 χώρες που εκπροσωπούνται στην Ένωσή μας είναι μεγάλη έκταση για μια τόσο καινούρια ένωση, ένα τόσο καινούριο σύνδεσμο. Πάμε από την Νορβηγία, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, στην Αγγλία, την Ιρλανδία και τον Νότο, τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία που σύντομα θα προσχωρήσει στο δίκτυό μας υπήρξαν πολλές συναντήσεις. Η Εσθονία, η Λουθουανία και η Δανία είναι κάποιες χώρες που ενδιαφέρονται και αυτές να μπουν στο δίκτυό μας. Έχουμε 3.200 παραγωγούς, ε, βιοτέχνες και παραγωγούς ε, χειροποίητου τυριού και γαλακτοκομικών προϊόντων που είναι άμεσα μέλη του δικτύου μας. Έχουμε διάφορες μορφές επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε. Οι άνθρωποι ε, που ζουν ε, ως ε, που παράγουν τυρί ως βιοτέχνες παίρνουν το, το γάλα και από τα δικά τους κοπάδια αλλά και από άλλα. οι υπόλοιποι που κάνουν χειροποίητο τυρί είναι το τυρί αυτό από γάλα και δικό, κυρίως ε, που αγοράζουν από γειτονικά αγροκτήματα. Το γάλα είναι κατσικίσιο, γελαδινό και τα λοιπά. Πρόκειται για οικογενειακές κυρίως επιχειρήσεις μικρής κλίμακας ε, που εργάζονται τοπικά σε επίπεδο τουλάχιστον προμήθειας ε, πρώτων υλών και χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους. Είναι οικογενειακές λοιπόν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Πρέπει βέβαια να επιμείνουμε στο γεγονός ότι ο τρόπος παραγωγής που ακολουθούμε και η αλυσίδα αυτή που έχουμε εμείς είναι ε, κάτι που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα που ε, εκπροσωπούμε, διότι όλο και περισσότεροι οι καταναλωτές ζητούν τα ντόπια προϊόντα, ζητούν ποιότητα, ε, οπότε ζητούν πληροφορίες σχετικά με το πότε και πού παρήχθη ένα προϊόν. Είναι λοιπόν ευρωπαϊκή τάση, αλλά και παγκόσμια ταυτόχρονα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή με το δίκτυο που έχουμε εκπροσωπούμε περίπου 40.000 επιχειρήσεις ε, του τύπου μας. Επειδή ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε εργατικά χέρια. Εκπροσωπούμε περίπου 100.000 θέσει εργασία. Μιλάμε για ανθρώπους ε, που ζουν ε, και εργάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο και οι οποίοι η οποία κατάσταση φθήνει σιγά σιγά, αλλά υπάρχουν και νέες δραστηριότητες. Είμαστε δυναμικοί λοιπόν. Έχουμε ανθρώπους στο δίκτυό μας που είναι αυτόνομοι και να το πούμε Γενικότερα δεν έχουν πάρει και τόσες επιδοτήσεις γεωργικές σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Να σας πω ποιο είναι το σύστημα πώλησης που έχουμε. Παραδοσιακά εμείς η παραγωγή, τουλάχιστον η παραγωγή ντόπιων προϊόντων, ε, πουλάμε είτε στο αγρόκτημά μας, είτε στο χωριό μας, είτε στην περιοχή μας. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σύστημα πώληση το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε πιο κατανοητό γιατί αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οι διοικητικοί ας πούμε δεν γίνονται κατανοητοί από τους διανομής οι οποίοι είναι τα εστιατόρια, τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι ειδικοί στο κτίρι. Είναι ένα μεγάλο λοιπόν σύστημα πώλησης, διευρυμένο και κυρίως μέσα από χονδρέμπορους περνάμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς ζούμε σε περιοχές λιγότερο πυκνοκατοικημένες για να βρει κανείς ε, πελάτες πρέπει να πάει στην πόλη. Οπότε μέσω από χονδρέμπορου προσπαθούμε να περάσουμε στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια και στα ειδικά μαγαζιά που πουλάνε τυρί. Κάποιε φορές εξάγουμε κιόλα. Παραγούμε με τον παραδοσιακό τρόπο, πολύ συχνά, με ε, γάλα, ε, ε, είναι παραδοσιακές οι μέθοδοι. Εδώ βλέπετε ακριβώς ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένα βαρέλια από ε, ξύλο. Μπορεί να έχουμε και κάποια εφασμάτινα ε, δοχεία ή από δέρμα. Είναι παραδοσιακές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για να πήξουμε το τυρί. Έχουμε αποστερεί το τυρί και παραδοσιακούς τρόπους ε, για να ε, πήξει κανείς και να παράγει το τυρί, να οριμάσει το τυρί. Η, παρουσία, η δραστηριότητά μας, όπως σας είπα, απαιτεί πολλά χέρια εργασίας, πολλά εργατικά χέρια. Οπότε, να σας πω ποιοι είμαστε εμείς. Είμαστε παραδοσιακή παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα ε, είμαστε και ικανοί, δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά αυτό που κάνουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας αφορά η υγειονομική ασφάλεια. Ξέρουμε πώς ε, να παράγουμε, ξέρουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε, γιατί χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια. Όπως ε, βλέπετε και από το μέσο του οδηγού, Γενικά θέλουμε να τηρούμε τις υγειονομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Δεν θέλουμε παρακλήσεις ως προς τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θέλουμε όμως μια προσαρμογή και μια ευελιξία. Γιατί δημιουργήσαμε το δίκτυο αυτό. Φαίνεται ότι παγκοσμίω ε, φαίνεται ότι γενικά το ευρωπαϊκό δίκτυο μας βοηθά να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας. Όταν αρχίσαμε να συναντιόμαστε με διάφορους ε, ευρωπαίους παραγωγούς και ενώσεις, γρήγορα καταλάβαμε ότι είχαμε κοινά προβλήματα. Οι περισσότερες ε, διοικήσεις ε, δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ουσία. Συνεχώς ε, μας επέβαλαν ρυθμιστικά άχθη, ε, γενικά δυσκολίες ε, σχετικά με το επάγγελμά μας, με τη δουλειά μας. Έπρεπε να κάνουμε καταγραφή και γενικά προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα σε εμά που είμαστε μικροί Πράγματα που κανονικά θα κάνουν, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πράγματα που μας ε, κάνουν να χρονοτριβούμε. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι και έχουμε και τα κοινά προβλήματα που μας ενώνανε. Το πιο σημαντικό στις δραστηριότητες μας σήμερα λοιπόν είναι η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση του τομέα μας, του κλάδου μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή η παραγωγή σε τοπικό επίπεδο, χειροποίητου του τυριού. Θέλουμε να κάνουμε lobbying σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης θέλουμε να κάνουμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων για την υγιεινή τις νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και το μάρκετινγκ, την τεχνολογία παραγωγής τυριού και γαλακτοκομικών προϊόντων. Υπάρχει ένα δίκτυο με ένα σύστημα ίντερνετ, ένα σύστημα δεδομένων που ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Και συναντιόμαστε κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό του τι έχει γίνει και της δουλειάς που κάνουμε έναντι της διοίκησης. Βασικά η περάσπιση των προϊόντων μας, η εκπροσώπηση του κλάδου, η αναγνώριση αυτής της μορφής παραγωγής είναι το πιο σημαντικό θέμα για μας. Γενικά μένουμε πάντοτε σε επιφυλακή σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να μας ε, προκύψουν ε, κάποιες, ε, κάποια ερωτήματα που προκύπτουν για το απαστερίο των τυρί και την ασφάλειά του. Προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τέλος πάντων τις μεθόδους μας. Προσπαθούμε δηλαδή να δείξουμε πώς λειτουργούν οι παραδοσιακοί παραγωγοί. Επίσης, θέλουμε να τοποθετηθούμε επί του γεγονότος ότι πολύ συχνά ε, μας βλέπουν ως ε, ε, διαφορετικούς γιατί απλώς πουλάμε σε τοπικό επίπεδο ή κάνουμε άμεση πώληση στον καταναλωτή ενώ η διαφορά μας είναι ο τρόπος παραγωγής. Ε, υπάρχουν ζητήματα διατροφικά, η σήμανση της προέλευσης του γάλατος. υπαρχουν ε, ζητηματα διατροφικα η σημανση της προελευσης του γαλατος πρεπει και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και να το προσαρμόσουμε στον τρόπο εργασίας μας η χρήση παραδοσιακών εργαλείων μεν, αλλά και ευελιξία ως προς τον κανονισμό για την υγιεινή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εξετάζουμε το νέο κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους. Τι είναι ο οδηγός στα σύντομα είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους παραγωγούς ε, να διαχειριστούν καλύτερα τους υγειονομικούς κινδύνους ε, στα εργαστηριά τους. Αλλά προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να εξηγήσουμε και στους επιθεωρητές τι κάνουμε. Ένα πολύ καλό εργαλείο λοιπόν επιτρέπει να μειώσουμε τα προβλήματα που έχουμε στην επικοινωνία με τη διοίκηση. Γιατί το φτιάξαμε. Η νομοθεσία για την υγιεινή μιλά για την ευθύνη του παραγωγού, για την υποχρέωση συγκεκριμένου αποτελέσματος, θέτει στο προσκήνιο τις αρχές καλών πρακτικών ε, παραγωγής και γι' αυτό φτιάξαμε αυτό τον οδηγό της καλής ε, πρακτικής που βασίζεται σε αυτή την μέθοδο, την HCCP. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον ε, οδηγό καλών πρακτικών που είναι ενισχύ και έγκυρος γενικότερα και που απαντά στα προσδοκίες των εθνικών διοικητικών αρχών. Η νομοθεσία για την υγιεινή και συγκεκριμένα το πακέτο για την υγιεινή μας επιτρέπει μια προσαρμογή στον τρόπο παραγωγής που έχουμε παραδοσιακά, όμως υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα στα αγροκτήματα, στα τυροκομεία μας. Κάποιοι θέτουν ένα αμφιβόλο την ευθύνη του παραγωγού και το, το αποτέλεσμα όπως ορίζονται στην νομοθεσία. Αυτά τα δύο στοιχεία καθώς ε, και η δυνατότητα χρήσης της ευελιξίας θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία μεν, όμως ε, στο πεδίο έχουμε σε κάποιες ε, χώρες τουλάχιστον προβλήματα με τη διοίκηση. Αν και η κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα. Πολλές από τις εθνικές ή περιφερειακές διοικήσεις μας έλεγαν δεν φταίμε εμείς που είναι αυστηροί κανονισμοί, είναι η Ευρώπη που φταίει. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτό τον Ευρωπαϊκό Οδηγό, ο οποίος ε, είναι επικυρωμένο σε επίπεδο ευρωπαϊκό και δεν μπορούν πια οι διοικήσεις να πούν ότι είναι το λάθος και το φταίξιμο στις Βρυξέλλες. Αυτοί φταίνε και αυτοί πρέπει να προσαρμοστούν. Η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι αυτή η καθεαυτή, μάλλον δεν είναι η νομοθεσία που δημιουργεί τα προβλήματα, αλλά ο τρόπος που εφαρμόζεται. Υπάρχει μια μορφή τυποποίησης των εργαλείων ευελιξίας. Κάποιοι επιθεωρητές δεν ξέρουν πολύ καλά πώς να γίνουν ευέλικτοι. Υπάρχει λοιπόν διαφορά σε επίπεδο εφαρμογής μεταξύ χωρών μελών. Για να το πω απλά, κάποιοι επιθεωρητές δεν έκαναν αποδεκτή τη νέα προσέγγιση της ευελιξίας. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί μεγάλη μάχη. Υπάρχει αυτή η τάση να μας λένε ότι μας αρέσει ο τρόπος που παράγεται, είστε χαρακτηριστικό στοιχείο της παράδοσης, ε, όμως θα σας βάλουμε σε καθεστώς εξαίρεσης. Όχι, δεν θέλουμε να είμαστε η εξαίρεση, θέλουμε να είμαστε πλήρως αναγνωρισμένοι. Η ευελιξία στον οδηγό. Έχω ήδη πει πολλά επί αυτού. Στην ουσία, ο οδηγός επιτρέπει να δοθούν παραδείγματα ευελιξίας που χρησιμοποιούνται σε διάφορα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την ευελιξία με τη χρήση του εξήλου, των φυσικών ε, χώρων ορίμανσης, ε, με τον έλεγχο των αντιβιωτικών. Όλα αυτά ε, δίνονται μέσα από τον οδηγό για να μπορούν ε, τα διοικητικά όργανα να τα χρησιμοποιούν. για να μπορούν ε, μέσα από αυτό τον οδηγό να λένε ότι όντως εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Το πρόβλημα της ευελιξίας βέβαια είναι ότι η εφαρμογή της ευελιξίας εξαρτάται από τη θέληση των κρατών μελών. Κάθε φορά εμείς λέμε ότι ναι, είμαστε υπέρ της ευελιξίας, αλλά είναι επιλογή του κράθε, κράτους μέλους πώς θα την εφαρμόσει και δεν εφαρμόζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. reconnaissance de, de, de de nos productions traditionnelles. Donc euh, ε, Ο οδηγός, όπως σας είπα, έχει επικυρωθεί. Είναι πλήρως ε, επικυρωμένος και γι' αυτό τον τρόπο, λόγο είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι ένα απλό εργαλείο για τους παραγωγούς για να μπορούν να κάνουν τις αναλύσεις τους και τους υγειονομικούς τους ελέγχους είναι ένα απλό εργαλείο που το αποδέχονται και η παραγωγή αλλά και η διοίκηση που γενικά είναι λίγο πιο συγκεκριμένη στην ερμηνεία της. Αυτός ε, ο οδηγός, ε, λοιπόν, επειδή είναι πρακτικός, ε, θα διδαχθεί. Έχουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που ονομάζεται Teach Easy και αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να ε, καταρτήσουμε τους παραγωγούς. Έχουμε τις εξαιρέσεις και τις προσαρμογές στον κανόνα. Εδώ έχουμε συστάσεις στον οδηγό, αλλά δεν έχουμε μια πλήρη επικύρωση. Ως προς την ευελιξία είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Τι θα κάνουμε στο εξής. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε. Σήμερα το πρωί μόλις είχαμε μία συνάντηση με την DG Sante και εκπροσώπους των εθνικών αρχών για να γίνει ένας ε, διάλογος με τις ελεγκτικές αρχές τους παραγωγούς τις οργανώσεις των παραγωγών η διοίκηση σε εθνικό, τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς θέλουμε αυτός ο οδηγός να υιοθετηθεί και να χρησιμοποιείται στην κατάρτιση των επιθεωρητών, των ελεγκτών. Το Tuning for Safer Food είναι μία από τις πρακτικές που έχουμε ενσωματώσει στον οδηγό. Θα έχουμε καλύτερη ε, κατάρτιση για τους παραγωγούς όπως σας είπα με το τι τσίζει και επίσης οι ίδιοι οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν δίκτυα που θα τους επιτρέπουν κάθε φορά που έχουν πρόβλημα να απευθύνονται στους ειδικού τεχνικούς που θα τους ταλύνουν. Θέλουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστήριξη γι' αυτό. Έτσι λοιπόν για, όλα αυτά, για όλους αυτούς τους λόγους ο οδηγός ήταν μια βάση και ένα πρώτο βήμα. Γενικότερα τώρα, και αυτό είναι η κατάληξη της ομιλίας μου, να πω ότι τα προβλήματα που παραμένουν τα έχω ήδη πει, αλλά θα επιμείνω έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της ευελιξίας η οποία δεν εξαρτάται πάντα από εμάς εξαρτάται από την καλή θέληση των κρατών μελών. Υπάρχουν στρεβλώσεις σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται οι παραγωγή στη μία χώρα και πώς σε άλλη. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν οι διευκολύνσεις που δίνονται σε μία χώρα να υφίστανται και να ισχύουν και στις άλλες. Βάσει των αποτελεσμάτων μας, δηλαδή των προϊόντων μας, ε, ε, Κάποιοι μπορεί να λένε ότι αυτά τα προϊόντα είναι λιγότερο ασφαλή από άλλα, αλλά δεν υπάρχει επιστημονική επικύρωση αυτού του ισχυρισμού. Έχουμε φτιάξει λοιπόν τον οδηγό, βελτιώνουμε τις υγειονομικές πρακτικές που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ευελιξίας. Είναι ένα ε, πρόβλημα που απομένει και θα θέλαμε η Ευρώπη να μας υποστηρίξει. Επίσης, ε, μόνο 15 είναι οι χώρες από τις 28 που συμμετέχουν στο δίκτυό μας. Δεν είναι πλήρης ο χάρτης, λοιπόν. Είναι δύσκολο να έχουμε νέες χώρες. Κάποιες φορές γιατί είναι πολύ απομονωμένη η παραγωγή και δεν είναι οργανωμένη. Αυτή η καλύτερη ε, δομή και διάρθρωση είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς παίρνει χρόνο. Και τέλος, το σημαντικό είναι να δείξουμε στη διοίκηση εθνική ή ευρωπαϊκή ότι οι εδετεραιότητές μας δεν έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εμπορευόμαστε τα προϊόντα μας, αλλά με τον τρόπο που τα παράγουμε. Για την θρεπτική αξία των προϊόντων και τη σήμανση, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να πω ποια είναι η θρεπτική αξία του τυριού μου. Όχι γιατί πουλώ άμεσα ή μέσω ενός εθνικού ενδιάμεσου, αλλά επειδή κατά τη διάρκεια του χρόνου το γάλα μου είναι διαφορετικό. Κάθε μήνα αλλάζει και τα χαρακτηριστικά του τυριού αλλάζουν. Αλλά και επειδή χρησιμοποιώ παραδοσιακές ε, μεθόδους ε, χειροκίνητες ε, με ξύρανση η οποία δεν είναι πάντοτε η ίδια. Δεν μπορώ να πω ποια είναι η θρεπτική αξία του προϊόντος μου. Δεν μπορώ λοιπόν να αναλύω συχνά την θρεπτική αξία και να αλλάζω και τόσο συχνά τις ετικέτες. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν και γι' αυτό και φτιάξαμε και κανόνες σε σχέση με την εμπορευματοποίηση αυτών των προϊόντων. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα πρόβλημα σημαντικό για το δικό μας τομέα δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ. Bene, grazie, veramente molto interessante. Ευχαριστώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Συγχαρητήρια για τη δημιουργία αυτού του δικτύου και για τη δουλειά που κάνετε. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Έχουμε διάφορου συναδέλφου που ζήτησαν το λόγο. Πριν από όλου, ο Ζωζέ Μποβέ που δεν τον βλέπω εδώ, αλλά ξεκινάμε με τον Ενρή Καντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. συγκινούμε με αυτή την παρουσίαση γιατί αν είναι σωστές οι πληροφορίες είναι σωστές που έχω είναι μια πιλωτική πρωτοβουλία πρόκειται για τον Στεφάν Λεφόλου που ξεκίνησε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε αυτό τον οδηγό για, για τις καλές πρακτικές Είναι μια επιτυχία. Το είπατε κι εσείς με τα λόγια σας. Για άλλη μια φορά, τη στιγμή που γίνεται πολύ λόγος για μια ανταγωνιστική γεωργία, δείχνεται, αποδεικνύεται ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη μέσα στη διαφορά τη. Και αυτό δείχνει ότι η ποικιλομορφία της γεωργίας είναι παρούσα και η γεωργία την οποία εσείς ε, προωθείτε είναι το ίδιο ανταγωνιστική με άλλα μοντέλα. Αυτό μας κάνει να διερωτηθούμε. Και αυτά που είπατε τα συνδέω με αυτά που είπαμε σήμερα το πρωί για μια έκθεση που ανέλαβε η συνάδελφος Ερένας Γαρσία για την παραγωγή βόηου όλου κρέατος. Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις και οι περιφέρειές μας έχουν διαφορετική ε, ιστορία και πολλές φορές η δραστηριότητα που μας είπατε εσείς ε, γίνεται ε, σε δύσκολες περιοχές, σε ορεινές περιοχές. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσει κανείς τη ζωή εκεί και μάλιστα εσείς το καταφέρνετε και με ανταγωνιστικό τρόπο. Δεν μπορούμε να μην το ακούσουμε αυτό. Με πρωτοβουλίες όπως αυτή που μας παρουσιάζετε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη μεγάλη ε, ποικιλομορφία που οδηγεί στην ισορροπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και το αίτημά σας για λογική. Και πιστεύω και εσείς το, το αποδεικνύετε ότι θα πρέπει να συνοδεύσουμε αυτές τις ε, θετικές πρωτοβουλίες και να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθούν αυτές οι δεστιότητες. Μπράβο σας, ευχαριστώ. Με καθησυχάζετε σίγουρα ορισμένους από εμά γιατί αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κακή ή καλή δραστηριότητα. Είναι αυτή η δραστηριότητα που επιτρέπει τη διαβίωση σε διάφορα μέρη με ιδιαιτερότητες. Για κάθε μια από τις εκμεταλλεύσεις μάλιστα. Έχουμε ας πούμε το πελαντών και το άμπρο του ροκαμαντούρ που είναι δύο διαφορετικά τυριά με καθόλου ίδια τρόπο παραγωγής, με εξαιρετική ποιότητα και με ε, τρόπο εκτροφής τελείως διαφορετικό. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ερικ. Επανήλθε ο Ζωζέ Μποβέ και έχει το λόγο. Oui, uh, bonjour. Ευχαριστώ και καλημέρα. Καλησπέρα. Χρήσιμο θα ήταν πόσο θα ήθελα πριν 40 χρόνια να τον είχαμε αυτόν τον οδηγό. Ανταυτού είχα τις διάφορες υπηρεσίες στην πλάτη μου που μου ζητούσαν να ακολουθήσω διαδικασίες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που έκανε, έκανε εγώ στη γεωργική μου στην κτηνοτροφική μου εκμετάλλευση. Ε, ασχολούμουν με τον αγροτοσυνδικαλισμό και έτσι με άφησαν κάπως ήσυχο. Αλλά επί χρόνια η γαλακτοκόμοι, κτηνοτρόφοι έχουν υποφέρει από αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες γιατί τους ζητούν ε, να ακολουθήσουν διαδικασίες τις οποίες δεν μπορούν να ε, φροντίσουν, να, να, να, να αναλάβουν ούτε για οικονομικούς λόγους ούτε εξαιτία της φύσεως του επαγγελματό τους, της, της δουλειάς τους. Υπάρχει λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό σε αυτόν τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών που είναι ότι δεν έχει νόημα να ζητούμε από αυτούς τους γαλακτοπαραγωγούς να ακολουθούν κανόνες σαν να τους λέμε ότι μόνο έτσι μπορείτε να περάγετε προϊόντα ασφαλή Ανταυτού καλύτερα είναι να ακούσουμε αυτούς τους παραγωγούς που ξέρουν τις παραδοσιακές δικασίες παραγωγής. Για μια φορά και επιτέλους ελήφθη υπόψη ε, η, αυτά που λένε οι ίδιοι οι και πιστεύω ότι το γεγονός ότι αυτές οι μέθοδοι παραγωγής γίνονται πλέον αποδεκτές σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό είναι εξαιρετικό και που αυτές οι, παρα... οι μέθοδοι παραγωγής πλέον χρησιμοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και επίσης κάτι ακόμα που θα ήθελα να χαιρετήσω είναι η πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε. Ήταν ε, ε, μια πρωτοβουλία την οποία υποστήριξαν πολλοί ευρωβουλευτές και ε, ένα άνθρωπο που νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε γιατί έμεινε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας ε, ο οποίος είναι ο κύριος Μισελ Ντουπό ε, ήταν, εργαζόταν ως βοηθός μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνταξιοδοτήθηκε. Πιστεύω ότι ο Μισελ Ντουπό συνέβαλε ε, σε, με κρίσιμο τρόπο τα μάλα σε αυτή την προσπάθεια. Tout à fait. Σα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, πρόκειται για μια πρωτοβουλία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους πρασίνους που έφεραν ε, το ευρωπαϊκό δίκτυο, στο ευρωπαϊκό δίκτυο αυτή την ε, ε, βιοτεχνική ε, εταιρεία, εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανταλουσίας ξέρω πόσες δυσκολίες έχουν αυτοί οι μικροί βιοτέχνες, μικρές εταιρείες που δίνουν μεγάλη αξία στην παραγωγή τους. Και όπως είπε και ο κύριος Μποβέ και ο κύριος Άντρου, είναι μια καταπληκτική ιδέα και νέο και ήδη αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει τις καλές πρακτικές και όπως είπε ο κ. Βοβέ ήδη αν τα ξέραμε Αυτά θα ήταν πάρα πολύ καλό αν υπήρχαν όλες αυτές οι καλές πρακτικές πριν από κάποια χρόνια όταν εμείς ξεκινούσαμε. Θέλω να χαιρετήσω εδώ και μία συγχωριανή μου από τη Γρανάδα, την ωραιότερη πόλη του κόσμου, λέμε μεταξύ μας και τη Μαρία Χεσού και Χιμένες και εκείνη θέλω να την καλωσορίσω καθώς και όλους τους συνοδεύουν. Καλωσορίσατε εδώ στις Βρυξέλλες ε, για να παρουσιάσετε και εσείς τη δική σας προσπάθεια. Πέρα από το να σας συγχαρώ για την εργασία σας και τη σημασία που έχει για τις ε, ε, μικρές, τα μικρά μέρη, τα μικρά χωριά Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μένουν στο μέρος τους, θέλουν να φτιάξουν μια δραστηριότητα για να κερδίζουν τη ζωή τους, να κάνουν, δώσουν και να δημιουργήσουν και μια θέση απασχόλησης. Δύο, ε, δεν είναι μόνο η αξία των θέσεων απασχόλησης, αλλά είναι και η αξία της συνοχής ε, του χώρου, κοινωνική αξία. θα είχαμε λιγότερη απερίμωση των ε, ε, περιοχών της υπαίθρου αν γίνονταν περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες. Γι' αυτό και θέλω να τη χαιρετήσω. Πιστεύω πως είναι πρωτοπόρα, πρωτοπόρο αυτό το δίκτυο. Ξέρω ε, και κάποιο άλλο δίκτυο βιοτεχνών. Πιστεύω πως είναι πρόοδος εδώ Η Γαλλία ξεκίνησε αυτή τη ε, διαδικασία. Εμείς έχουμε αντιγράψει πολλά από αυτά που γίνονται στη Γαλλία. Και πρέπει να βελτιώσουμε τις ηθίκες διαβίωσης των ανθρώπων. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί ε, η υγειονομική ε, ε, επιθεώρηση βάζει το ίδιο καλάθι το, ε, αυτόν τον παραγωγό που φτιάχνει 30 κεφάλι τρίτη την ημέρα με αυτόν που φτιάχνει 300 ή 3.000. Μα δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό είδος προϊόντος. Και αυτή τη διαφορά πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία των καλών πρακτικών και την προσαρμογή αυτών των ευρωπαϊκών ε, ρυθμίσεων, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Όχι μόνο για το τυρί, αλλά πιστεύω πως αυτό αποτελεί ένα προηγούμενο. Είναι ένα προηγούμενο και για τα υπόλοιπα προϊόντα. Και η επιτυχία είναι μεγάλη. Σας συγχαίρω για αυτή τη δουλειά. Εμένα αυτό που με ανησυχεί επίσης είναι η χρήση της λέξης artisanal, δηλαδή τεχνικός, παραδοσιακός και ε, artisanal. Είναι, ένα, είναι μια σήμαση που φέρουν και προϊόντα τα οποία παράγονται βιομηχανικά. Ε, ως καταναλωτές ε, θα πρέπει να προσέχουμε. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές οι ετικέτες για προϊόντα τα οποία δεν είναι βιοτεχνικού τύπου είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε σύγχυση του καταναλωτή. γιατί ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει συγκεκριμένη τιμή για ένα προϊόν που ξέρει ότι φτιάχνεται ε, ε, παραδοσιακά και βιοτεχνικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κλάρα και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Μπούντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον φίλο και συνάδελφο από το δίκτυο ε, που μας παρουσίασε αυτή, τον οδηγό βελτίστων πρακτικών. Τέτοιου οδηγούς βελτίστων πρακτικών θα θέλαμε και για πολλούς άλλους τομείς, όχι μόνο για τα γαλακτοκομικά. Μαζί με τον φίλο και συνάδελφο Νταντά ε, επισκεφτήκαμε την Γαλλία, το Βέλγιο, την Αυστρία και είδαμε γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και διαπιστώνω ότι πολλοί ε, πολίτες τα επιθυμούν αυτά τα μικρά γαλακτοκομεία στις τοπικές τους περιοχές. Στη Ρουμανία έκλεισαν πολλά γιατί δεν αντιλαμβανόταν ο κόσμος γιατί να χρειάζονται ε, και τι ακριβώς προσθέτουν, τι πιάνει προσθέμενη αξία. Δυστυχώς, πολλές φορές οι ελεγκτέ επιβάλλουν κυρώσει μετά από έλεγχο χωρί κανείς να έχει καταλάβει ποιο ήταν το πρόβλημα σε αυτή την μονάδα παραγωγής και πρόκειται για ελεγκτές οι οποίοι πολλέ φορέ ε, αντιμετωπίζουν το ζήτημα θεωρητικά χωρίς να έχουν και οι ίδιοι μια εμπειρία από ένα αγρόκτημα από μια μονάδα παραγωγής. Σα υποστηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να σα υποστηρίζουμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας δίνετε τη δυνατότητα να σας υποστηρίζουμε με τις πρωτοβουλίες σας, γιατί πραγματικά εμεί θέλουμε να, να, να υποστηρίξουμε τέτοιες ε, μικρές εκμεταλλεύσεις. Το ερώτημα που θα ήθελα να σα θέσω, είναι το εξή. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μεταξύ σα, μέσω του δικτύου δηλαδή, ε, κάποιο, κάποιο σύστημα διανομή, κάποια σημεία πώληση. Έτσι ώστε να απευθυνθείτε σε καταναλωτές σε περισσότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Και κάτι ακόμα, δεν είδα τη Ρουμανία να εμφανίζεται με μπλε στο χάρτη σας. Έχετε επικοινωνήσει με κάποιους παραγωγούς από τη Ρουμανία. Τι γίνεται με τη χώρα μου. E, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συγχαίρω και εγώ τον προσκεκλημένο μας για τις πρωτοβουλίες του δικτύου του και τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών. Γνωρίζουμε ο γαλακτοκομικός τομέας περνάει μια κρίση και αυτό έχει πλήξει όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχουν πληγεί ιδιαίτερα και ακόμα περισσότερο τα νέα ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη δηλαδή. Στην Κροατία ο αριθμός των γαλακτοπαραγωγών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 60%. Την τελευταίο χρόνο μόνο αυξήθηκαν οι εισαγωγές γάλακτος προς την Κροατία 281% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα που είχαμε το 2012. Αυτό σας δείχνει για πόσο μεγάλη είναι η κρίση του τομέα ε, των γαλακτοκομικών στην Κροατία. Επομένω, χρειάζεται να βρούμε άλλων ειδών λύσει γιατί οι τωρινέ δεν, δεν λειτουργούν. Μιλήσατε για την αυτοργάνωση των ε, γαλακτοπαραγωγών και συμφωνώ. Και το ερώτημα μου προς εσάς είναι εσείς πώς τα καταφέρατε και τι θα μπορούσατε να προτείνετε σε άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν προς στιγμή τέτοια δίκτυα. Πώς μπορούν να οργανώσουν τους παραγωγούς και να δημιουργήσουν τέτοια δίκτυα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε με νομοθετικά μέτρα να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τι περιμένετε από εμάς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ή μήπως χρειάζονται κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες αλλαγές στους υφιστάμενους κανονισμούς. Σας ευχαριστώ. Σέρβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ για να μας παρουσιάσετε αυτό τον οδηγό καλό πρακτικών γιατί εγώ από τα όσα άκουσα πιστεύω πως υπάρχει πολλοί κόσμος που βρίσκεται σε αυτή την Επιτροπή και που μας έχει τύχει να ζήσουμε από διαφορετικές προοπτικές αλλά κάποιο είδος επαφής είχαμε για να δώσουμε αξία και για να διατηρηθούν τα γεωργικά προϊόντα, τα... οι μικρές εκμεταλλεύσεις, η άμεση ε, πώληση και επίσης θα ήθελα να γνωρίζω τι, ποια βήματα περισσότερο θα πρέπει να κάνουν οι ε, διοικητικοί μηχανισμοί αλλά και η και το Ευρωκοινοβούλιο για να συμβάλλουμε ώστε αυτή αυτή, αυτός ο οδηγός, αυτοί οι κανόνες να εφαρμοστούν με σωστό τρόπο ή να μπορέσουν όλοι μέσα στο Ευρωπαϊκή Επικράτεια να προχωρήσουν. Και δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω τι συγκεκριμένες προτάσεις έχετε για τη σήμανση, για την ετικετοθεσία. Θέλετε να γίνει κάποια διαφορετική ετικετοθεσία, διαφορετική σήμανση. Πώς να το δουλέψουμε γι' αυτό ώστε να μην υπάρξουν δυσκολίες και έπειτα προς τους ευρωβουλευτές που σήμερα είμαστε εδώ. Θεωρώ ότι από όλε τις πολιτικές ομάδες χαιρετήσαμε αυτή, αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα να αναλάβουμε την ευθύνη να σκεφτούμε συλλογικά για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Πριν, ε, Κλάρα, εσύ αναφέρθηκες ε, σε αυτό που σε ανησυχεί και που και εμένα με έχει ανησυχήσει από την συνδικαλιστική ε, προπτική ε, που ήμουν προηγούμενα, που δούλευα με όλα αυτά και είναι σαφές ότι συχνά η παραδοσιακή κατασκευή, η παραγωγή τυριού που έχουμε σε πολλά μέρη, πώς θα αποφύγουμε να πέσει στα χέρια των, ε, της μεγάλης βιομηχανίας. Είναι πολύ σαφής ευθύνη των ε, τοπικών αρχών και των αρχών εν γέννη, όταν δηλαδή κανείς νομοθετεί θα πρέπει να προσπαθήσει να εμποδίσει ο ορισμός αυτός να μην πέσει στα χέρια των μεγάλων βιομηχανιών. Στη Γαλλικία είχαμε έναν αγώνα αρκετά σημαντικό για να εμποδίσουμε ακριβώς ε, η ονομασία του η ονομασία ε, παραδοσιακή παραγωγή ε, να πέσει στα χέρια της μεγάλης βιομηχανίας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Μεγάλη ευκαιρία να δούμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς στηρίζονται αυτές οι πρωτοβουλίες. Και τώρα θα σου δώσω το λόγο για να απαντήσεις και στις ερωτήσεις στους συναδέλφους που σου έθεσαν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι και εγώ είμαι πολύ συγκινημένος ε, γιατί και, πράγματι ξέχασα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ευρωβουλευτέ που μας βοήθησαν από την αρχή της πρωτοβουλία, ιδιαίτερα τους Γάλλους ευρωβουλευτέ, ε, αλλά και από την Πολωνία και από αλλού. Δεν θα μπορούσα να σας ευχαριστήσω όλους γιατί δεν έχω τον κατάλογο, αλλά πάντως ε, συνολικά να πω ότι σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Και πράγματι και εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Μισελ Τζουπό, ο οποίο πάντοτε ε, διευκόλυνε τι επικοινωνίε μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια και δεν είμαστε πάντα στι Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και η έπαιξε κρίσιμο ρόλο. Το ερώτημα που ετέθη ε, από ένα μέλος κοινοβουλίου κάποια στιγμή ήταν ε, πόσο έχουμε οργανώσει τους παραγωγούς και γιατί η Ρουμανία δεν εκπροσωπείται ακόμα και αυτό που είπατε ε, ότι πριν από 40 χρόνια ε, στη Γαλλία σας έπριζαν με ανόητους κανονισμούς. Να σας πω ότι δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα ακόμα. Ε, έχουμε συνεισφέρει σε μία αλλαγή. Έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε με χώρες, με παραγωγούς από χώρες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο δίκτυό μας, ανάμεσά τους η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Εστονία, η Δανία. Ε, άρα δεν είναι μόνο οι χώρες που είδατε στο χάρτη στη διαφάνεια. Ε, και ιδίω ε, το πρόβλημα της μη συμμετοχή το έχουμε με χώρες στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και αλλού. Επομένως, Προσπαθούμε να προσελκύσουμε ε, παραγωγούς και από εκεί. Πάντως το πρόβλημα της υπερβολικά αυστηρής εφαρμογής των κανονισμών παραμένει και είναι κάτι στο οποίο έρχομαι και επανέρχομαι. Ε, το ζήτημα είναι το εξής κατά την άποψή μου. Ο ίδιος ο κανονισμός ο ευρωπαϊκός επιτρέπει ε, ευέλικτη εφαρμογή του ή μια κάποια διακριτική ευχέρεια. Όμως τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που επιλέγουν τους συγκεκριμένους τη συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής και είναι εκείνα που έχουν επιλέξει να μην ε, είναι διαλλακτικά. Ε, από άγνοια, από ε, δυσκολία διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης. Για, για, για διάφορους λόγους έχουν επιλέξει να μην εφαρμόζουν αυτές τις ευέλικτες διατάσεις που τους δίνει ο κανονισμός. Γιατί ε, αυτό θα χρειαζόταν περισσότερη δουλειά τελικά. Θα χρειαζόταν μεγαλύτερη επαφή με τους παραγωγούς για να εξηγήσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους. Ε, έχουμε λοιπόν επαφές και με άλλους παραγωγούς στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία που θέλουν να ενταχθούν. Πάντως πρόκειται για χώρες στις οποίες δεν υπάρχει μια ε, καλά οργανωμένη δομή των επαγγελματιών παραγωγών. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Χρειάζεται χρόνος. Ε, το δίκτυό μας ε, εργάστηκε για την παραγωγή αυτού του οδηγού βέλτιστων πρακτικών και συμμετείχαν σε, αυτή, σε αυτό, στη σύνταξη αυτού του οδηγού και οι ίδιοι οι παραγωγοί ε, και όμως ε, ειδικοί, τεχνικοί που συνεργάζονταν με τους παραγωγούς με τη σειρά τους Το οποίο σημαίνει ότι για να ενταχθεί λοιπόν μια νέα χώρα για να... η οποία δεν είναι ακόμα στο δίκτυό μας θα πρέπει εμείς ε, η παραγωγή των μικρών εκμεταλλεύσεων μαζί με κάποιους τεχνολόγους τροφίμων ειδικού στο θέμα να επισκεφτούμε αυτές τις χώρες, να μιλήσουμε με τους παραγωγούς, να μιλήσουμε με τη δημόσια διοίκηση αυτών των χώρων, να τους εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί, να τους εξηγήσουμε πώς μπορούν να εφαρμόζουν πιο σωστά και πιο ευέλικτα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον κανονισμό στην, στην περίπτωση των μικρών παραγωγών. Αυτό λοιπόν χρειάζεται χρόνο και πόρους. Αυτή τη στιγμή το δίκτυό μας είναι μικρό ε, και για να το πω ευθέω, ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ουσιαστικά οικονομική βοήθεια. Ήταν ε, το ίδιο είδος βοήθεια που χρειαστήκαμε για να παραγάγουμε και αυτόν τον ε, οδηγό βέλτιση των πρακτικών. Πρόκειται για μια μικρή, ένα μικρό οργανισμό, μια μικρή οργάνωση. Χρειάζεται χρήματα. Για το ζήτημα τη τον, Το αίτημά μας είναι απλό. Υπάρχει ένα άρθρο στον κανονισμό το, για την ετικετοθεσία στα τρόφιμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε μικρές εκμεταλλεύσεις οι οποίες ακολουθούν παραδοσιακές πρακτικές να το λένε στην ετικέτα ε, αυτό μας διευκολύνει και προσθέτουμε το ότι θα πρέπει να γίνεται η, η πώληση είτε τοπικά ή μέσω ενός ε, ενδιάμεσου. Εμείς θα Έλαμε ε, να προσθεθεί μάλλον όχι, να, να, να μην υπάρχει αυτή, η διατύπωση η οποία περιορίζει τις πωλήσει μας στον τόπο παραγωγής. Φανταστείτε την δική μου περίπτωση, Γον Αλπ γίνεται η παραγωγή στην περιοχή της Λιών, υπάρχουν πιθανοί πελάτες στο Παρίσι, ε, ε, ε, ε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια ετικέτα η οποία να βιοθέτει τα θρεπτική αξία του προϊόντος μου και να το πωλήσω στο Παρίσι λέγοντας ότι είναι τοπικό, ότι είναι παραγωγή παραδοσιακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει στα κράτη-μέλη να δείξουν τη διαλλακτικότητα ή τη διακριτική ευχαίρεια από τους επιτρέπει ο αυτό που ανταπαντούμε θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός δικτύου στο οποίο να συμμετέχουν η παραγωγή αφενός με εκπροσωπούμενοι από οργανώσεις όπως η δική μας και οι ελεγκτές, τα φορείς ελέγχου των κρατών μελών, έτσι ώστε να συζητούν τα προβλήματα εφαρμογής του κανονισμού στην πράξη και να δείχνουν και να συζητούν ε, ε, πώς μπορεί να επιδεικνύεται αυτή η διαλλακτικότητα. Εάν έχουμε ένα δίκτυο στο οποίο θα έρχονται από τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη, οι φορείς ελέγχου, οι ελεγκτές. Υπάρχουν κάποια κράτη που έχουν μείνει πιο πίσω στην εφαρμογή αυτής της ε, διακριτικής ευχέρειας και πιστεύω ότι θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς αυτά τα κράτη-μέλη ότι είναι επιθυμητή αυτή η διαλλακτικότητα, αυτή η ευελιξία. Νομίζω μέχρι εδώ μπορώ να ε, μιλήσω εγώ. Ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την τοπική παραγωγή και μια, ε, τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη. Ε, γνωρίζουμε, ακριβώς προσπαθώντας να ενισχύσουμε την διαφορετικότητα πρέπει να γνωρίσουμε ότι έχουμε διαφορετικές νοτροπίες. Δεν μιλούμε όλοι αγγλικά και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που κατάφεραν, καταφέραμε όλοι μαζί με τη βοήθεια όλων να καταλήξουμε σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα που σας παρουσιάζω σήμερα. Felicidades. Felicidades. De nuevo, eh, Εξ ονόματος της Επιτροπής και όλων των Ευρωβουλευτών Σα συγχαίρουμε για τη δουλειά που κάνετε εσείς ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου και όλοι όσοι ε, εργάζονται καθένας ε, στην δική του περιφέρεια για αυτή τη σπουδαία δουλειά. Τώρα, ολοκληρώσαμε την εξέταση της ημερήσιας διάταξης που είχαμε για σήμερα. Έχουμε ε, να δοκιμάσουμε ε, τα τυριά που μας προσφέρει ε, στο τρίτο, στο τρίτο όροφο του, του άλλου κτηρίου του Γιάννα στις 6. Και επειδή τελειώσαμε λίγο νωρίτερα, στο Γιάννα λοιπόν. Να έρθετε όλοι. Αύριο στις 9 θα συνεχίσουμε με τον πρόεδρο και που αύριο θα είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια και στον κύριο Μποβέφ.